Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην πρώτη συνεδρίαση του 2020. Ε, Γνωρίζετε όλοι ότι Είμαστε σε μια καθοριστική στιγμή για τη γεωργική πολιτική, γιατί αφενός έχουμε το θέμα της ε, δημοσιονομικής ε, προοπτικής από το 21 μέχρι 27 και βεβαίως ε, κρίσιμο το έτος που διανύουμε και για το περιεχόμενο της γεωργικής πολιτικής, γιατί όσοι έχουν τώρα τα πράγματα και φέτος ε, θα κληθούμε να αποφασίσουμε για το τι πορεία θα ακολουθήσουμε για την πορεία 21 έως 27. Ως εκ τούτου η δική μας Επιτροπή βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινή γνώμης της Ευρώπης και αυτό όχι μόνο όσον αφορά τους γεωργούς αλλά και πάρα πολλούς άλλους. Έχουμε μία διευρυμένη πολύ ε, πληθωρική θα έλεγα η διάταξη και γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με τη μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει ε, για τα θέματα, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και θα ήθελα να σας ε, επισημάνω ότι και αυτή η συνάντηση μεταδίδεται μέσω διαδικτύου και η διερμηνία υπάρχει σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από εστονικά, λετονικά, μαλτέζικα και ε, κέλτικα. Πάμε λοιπόν στο σημείο υπαριθμών 3 της ημερήσιας διάταξης που είναι έγκριση των πρακτικών. Αν δεν έχετε αντίρρηση εγκρίνονται και τα πρακτικά. Και ως εκ τούτου περνάμε στο επόμενο θέμα, στο σημείο υπερθυμών 4 της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά στη συνεδρίασή μας την Υπουργό Γεωργίας της Κροατίας και την Προεδρεύουσα Μαρία Μπούκοβιτς. Θα ήθελα, Βούκοβιτς, ελπίζω να το, ε, να το πρόφερα σωστά. Σας καλωσορίζουμε κυρία Βούκοβιτς. Βούτσκοβιτς. Ξεκινάμε λοιπόν τη συνεδρίαση. Η ε, Κροατική Προεδρία έχει υπόψη να κάνει πάρα πολλά υπό το σύνθημα «Ισχυρή Ευρώπη, πάρα πολλές προκλήσεις». Πιο συγκεκριμένα όμως αυτό που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας είναι τι ακριβώς επιθυμείτε, και ε, πόσο ουσιαστικά θέλετε να προχωρήσετε στο θέμα της κοινή γεωργικής πολιτικής τόσο κατά το πρώτο εξάμεινο ε, όσο και στη συνέχεια. Ενδιαφέρουν και το θέμα των ε, δημοσιονομικών προοπτικών, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που είμαι σίγουρος ότι θα σας τα θέσουν οι συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ και τώρα πλέον έχετε τη δυνατότητα ε, για ένα τέταρτο, 15 περίπου λεπτά, να παρουσιάσετε τις απόψεις σας. Μετά θα ακολουθήσει συνεδρίαση ε, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις πρώτα από τους συντονιστές και μετά από όλους τους άλλους ε, συναδέλφους. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε Πρόεδρε της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριε Λίνς. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, κυρίε και κύριοι, νιώθω ιδιαίτερη τιμή για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω τι προτεραιότητε τη Κροατική Προεδρία στα θέματα γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και δασοκομεία. Η Κροατία αναλαμβάνει την Προεδρία σε μια πολύ δύσκολη στιγμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι έχουμε μια σειρά εκκρεμών και περίπλοκων πολιτικών θεμάτων. Για μα αυτό είναι μια πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα και τεράστια τιμή για μια χώρα που είναι το νεότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Προεδρία χωρίς καν να έχει πληρώσει 7 χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το σλόγγαν μας είναι «Η «Ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις» και έτσι με βάση και, τη στρατηγική, και το στρατηγικό θεματολόγιο 2019-2024 θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ κρίσιμες προκλήσεις όπως η άνηση ανάπτυξη οικονομική, οι κλιματικές αλλαγές, η μετανάστευση και η ασφάλεια. Τέσσερις είναι οι βασικές προτεραιότητες της Κροατικής Προεδρίας και πρώτη από αυτές είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες και τις προοπτικές όλων των Ευρωπαίων πολιτών με ισότιμη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Γι' αυτό όμως χρειαζόμαστε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό και μια γεωργία που θα κρατάει την εξέχουσα της θέση. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρει όχι μόνο τους γεωργούς και τους κατοίκους των αγροτικών περιοχών, αλλά όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό στη διάρκεια της κρατικής προεδρίας θα αναδείξουμε την σημασία που έχει η ανοιχτή επικοινωνία με τους ε, νομοθέτες. Εξού ε, και η σημερινή ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να συμβάλλουμε στη δημιουργία καλύτερων πολιτικών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ταυτόχρονα μία από τις πιο περίπλοκες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπτύσσεται σε πολλούς κύκλους ε, μεταρρυθμίσεων. Ε, βέβαια, οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διάπουν και τις επόμενες μεταρρυθμίσεις θα είναι κατά τη γνώμη της Προεδρίας η απλούστευση, επικουρικότητα και η βιωσιμότητα. Για πολλούς ε, λόγους ε, ε, εδώ και πολλά χρόνια συμπληρώσαμε το νομικό πλαίσιο της κοινή γεωρικής πολιτικής με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα μια σχετικά δυσνόητη και περίπλοκη και δύσκολη εφαρμογή γεωρική πολιτική. Μάλιστα πρόσφατα ήταν χαρακτηριστική μια δήλωση Γεωργού που είπε ότι θέλω να τηρήσω τους κανόνες, αλλά αλλάζουν τόσο συχνά που είμαι βέβαιος ότι κάπου έκανα λάθος. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πού ακριβώς έκανα αυτό το λάθος. Οπότε οποιαδήποτε προσπάθεια απλούστευσης ε, της κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής είναι ευπρόσδεκτη. Και αυτό θα προσπαθήσει η Κροατική Προεδρία να βελτιώσει, ε, να απλουστεύσει την κοινή γεωρική πολιτική και τους κανονισμούς, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στα πλαίσια του σχεδιασμού και των εφαρμοστικών μέτρων των εθνικών στρατηγικών ε, σχεδίων. Δεν θέλουμε υπερβολικά αυστηρές και δυσανάλογες κυρώσεις σε περίπτωση που έχουν ε, ε, πραγματοποιηθεί ακούσια σφάλματα. Ε, επίσης θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο επικείς και με τα κράτη-μέλη όταν ε, λόγω των ιδιαιτερότητων τους αποκλίνουν μερικέ φορές από την εφαρμογή των σχεδιασμένων μέτρων. Για λόγους όμως που διαφεύγουν το ελέγχου τους. Η κοινή γεωργική πολιτική θα συνεχίσει την αύξηση των αρμοδιοτήτων και ευθυνών των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των μέτρων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η, Ευρωπαϊκή, η Κροατική Προεδρία είναι υπέρ αυτής της προσέγγισης. Και λόγω των διαφορών και των διαφορετικών συνθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη είναι τα πιο αρμόδια να πούν πόσα και ποια μέτρα θα συμβάλλουν στην υλοποίηση των κοινών στόχων. Και ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες της ε, γεωργίας τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ευέλικτες λύσεις και κατά την επεξεργασία των εθνικών στρατηγικών σχεδίων. Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια για τη βιωσιμότητα που εδώ και πολλά χρόνια είναι η κατευθυντήρια γραμμή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και μάλιστα θα δώσουμε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 φιλοδοξιών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βέβαια, ένα εκρεμές ακόμη αλλά κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση αυτών των αυξημένων φιλοδοξιών. Η πρόταση των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει νέα μέτρα και πολύ πιο αυστηρές υποχρεώσεις των πολιτών, των γεωργών για την ε, ε, προστασία του κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε την αύξηση αυτών των κλιματικών δραστηριοτήτων, να ταυτόχρονα προτείνεται περικοπή του γεωργικού προϋπολογισμού. Η υλοποίηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών μας ε, στόχων και φιλοδοξιών ε, δεν θα καταστεί δυνατή αν δεν εξασφαλίσουμε αύξηση του προϋπολογισμού της κοινή γεωργικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της μελλοντικής πολιτικής, ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη της μέχρι τώρα πρόοδος της ΚΑΠ και να αναγνωρίσουμε τις σημαντικές προσπάθειες των γεωργών που έχουν επενδύσει στην παραγωγή τους και ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εδώ και χρόνια στόχος της κοινή γεωργικής πολιτικής δεν είναι μόνο η παραγωγή τροφίμων, αλλά όλο και περισσότερο έχουμε περιβαλλοντικές και κλιματικές πτυχές που στο πλαίσιο της κοινή γεωρικής πολιτικής ε, θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα και απαιτήσει για τους παραγωγούς. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τη γεωργία, να μην τη βλέπουμε ως πρόβλημα ή κίνδυνο για το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα. Οι γεωργοί στην Ευρώπη για πολλές γενιές ε, ζούσαν και εργαζόταν στον ίδιο χώρο και θέλουν να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν την ε, γη τους για να την κληροδοτήσουν σε επόμενες γενιές. Ενστικτοδός οι γεωργοί με ρίμνησαν για τη βιωσιμότητα πολύ πριν εμφανιστεί αυτός ο όρος στο πολιτικό μας λεξιλόγιο. Πέραν του μεταρρυθμιστικού πακέτου της κοινή γεωργικής πολιτικής, ε, ύψιστη προτεραιότητα της κρατικής προεδρίας θα είναι η έγκριση του κανονισμού για τις μεταβατικές διατάξεις για το 2021. Η πολιτική συζήτηση επί της προτάσεως αυτής θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλία. και στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο στους επόμενους τρει ή τέσσερι μήνες. Και καλούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί το συντομότερο τριμερής διάλογος, ώστε να προσδιορίσουμε το νομικό πλαίσιο και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καταβολή των ενισχύσεων στους γεωργούς κατά το 2021. Η Προεδρία ε, θεωρεί ότι με τις νομοθετικές πράξεις δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε πολιτικά συμφέροντα, αλλά να έχουμε υπόψη το συμφέρον των ε, ε, γεωργών. Θα πρέπει να περιοριστούμε σε συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο και με, τον, με την αρχή παλί, ε, παλί κανόνες και νέα μέσα θα πρέπει να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για να αποφύγουμε τον, επικίνδυνο, τον, τον κίνδυνο διακοπής της καταβολής των ενισχύσεων στη μεταβατική περίοδο. Επίσης, ε, πολύ σημαντικό για την κρατική Προεδρία είναι η Νέα Πράσινη Συμφωνία και η μελλοντική στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Βέβαια, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν πολύ θετικές για, τα, για τις προτάσεις αυτές, αλλά έχουν μείνει πολλές εκκρεμότητες και θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, κάτι που θα αποτελέσει προτεραιότητα και της Κροατικής Προεδρίας, ιδιαίτερα στα πλαίσια του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλίας. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε αλλάξει τρόπο σκέψης. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποδίδουν όλο και περισσότερη σημασία στη διαφύλαξη υγιούς, βιώσιμου και ποικίλου περιβάλλοντος με σκοπό να ε, διαφυλαχθεί και να κληροδοτηθεί και σε επόμενες γενιές. Και γι' αυτό στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εντάσσονται στο πλαίσιο μιας γενικής φιλοπεριβαλλοντικής προσέγγισης και θεωρώ ότι με φιλόδοξο και οραματικό τρόπο θα μας επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, βιώσιμο και καινοτόμο ευρωπαϊκό σύστημα τροφίμων. Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής έχουμε και τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο που θα συμπληρώσει τα ήδη υψηλά πρότυπά μας στη γεωργία και την παραγωγή των τροφίμων. Η Κροατική Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη περιορισμού της χρήσης φυτοφαρμάκων, που είναι σημαντικό για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Η Προεδρία μας ε, θα προωθήσει την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία και Εναλλακτικού μη χημικού φυσικού τρόπου καταπολέμηση των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, γιατί θέλουμε να περιορίσουμε τη χρήση και την εξάρτησή μα από χημικά φυτοφάρμακα. Ε, Χωρί όμω ταυτόχρονα να περιορίσουμε την ανταγωνιστικότητα τη γεωργίας μα. Πολύ σημαντικό θέμα είναι και η καλή μεταχείριση των ζώων, θέμα προσφυλές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και χαίρομαι που η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει το έργο της πλατφόρμας για την ευζοία. Και μάλιστα εμείς συμμετείχαμε στην πλατφόρμα αυτή από τη δημιουργία της και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Θέλουμε επικοδομητικό έργο ε, για τα θέματα καλής μεταχείρισης των ζώων, στην μεταφορά, την εκτροφή των ζώων και την ε, αποτροπή και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου κατοικιδίων ή ζώων συντροφιάς. Επίσης, ε, στα πλαίσια του, της Νέας Πράσινης Συμφωνίας θα ήθελα να αναφερθώ στο σημαντικό ρόλο της δασοκομείας οι, κράτες, οι χώρες μέλη εδώ και χρόνια ασχολούνται με την προστασία και την ανανέωση των δασών και παγκοσμίω. Και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δάση μετά το 2020. Την σχετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περιμένουμε ε, στο τρέχον έτος. Είναι σημαντικό ε, να προστατεύσουμε τα δάση γιατί προστατεύουν τη βιοπικιλότητα Φυσικά, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, γιατί το επίπεδο και το ποστό δασοκάλυψης στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε τη θέση μας παγκοσμίω και να προαγάγουμε μία αηφόρο διαχείριση δασών. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σημαντική οικονομική δύναμη και καταναλωτής προϊόντων από κάθε μέρος του κόσμου και ταυτόχρονα με την πλούσια εμπειρία της για την αηφόρο διαχείριση των δασών, πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην προστασία των δασών, ιδιαίτερα σε απειλούμενες περιοχές. Η Κροατία ασχολείται με την αηφόρο διαχείριση των δασών πάνω από 250 χρόνια και είναι αποδεδειγμένο ότι η αποτελεσματική διαχείριση των δασών μπορεί να εξασφαλίσει και ε, την διαφύλαξη των οικονομικών, οικολογικών και κοινωνικών λειτουργιών του δάσους προς όφελος ε, ολόκληρων κοινοτήτων. Στα πλαίσια αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον καλύτερο τρόπο αντίδρασης προκειμένου να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές και να επιταχύνουμε την προσαρμογή των δασικών συστημάτων στις νέες συνθήκες. Πολλές ε, προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας και πολύ σοβαρές, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολύ θετικά παραδείγματα που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε για την ανάπτυξη του τομέα. Οι νέες τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους φυσικούς πόρους και θα συμβάλλουν στην i4 και βιώσιμη παραγωγή. Επίσης θα διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών στην πληροφόρηση. Οι νέες τεχνολογίες ε, πιστεύω ότι θα καταστήσουν την γεωργία πιο ελκυστική και για τους νέους και θα τους κρατήσουν στις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε μια ηλικιακή ανανέωση στην ε, γεωργία και την καταπολέμηση της, ε, στη φυλήση της απερίμωσης της υπαίθρου, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλά Γι' αυτό θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες για την αναζήτηση νέων τεχνολογικών λύσεων. Επίσης θα προωθήσουμε την βιοοικονομία. Είναι έννοια που προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες και δυνατότητες σε τομείς όπως η γεωργία και η δασοκομεία. Η βιοοικονομία μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, να δημιουργήσει νέες ε, ευκαιρίες ε, επιχειρηματικότητας και θέσεις εργασίας και να καταλήξει σε παραγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω τον μεγάλο ρόλο και την ανάγκη αναγνώρισης της συμβολής των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Σε πολλές χώρες μέλη, οι μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οπότε θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την ε, δεσπόζουσα σε πολλές ε, χώρες, κυρίαρχη μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν ε, ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν και να προκόψουν και να ενισχύσουμε την θέση τους προκειμένου να ανανεώσουμε, να αναζωογονήσουμε τις αγροτικές μας περιοχές και τα χωριά μας και η, Ευρωπαϊκή, και η Κροατική Προεδρία αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν μπροστά τους ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εξάμεινο προκειμένου να συνεργαστούμε για να εξασφαλίσουμε ένα καλό νομικό πλαίσιο για τη μελλοντική κοινή γεωρική πολιτική. Προσβλέπω σε αγαστή συνεργασία και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση του προγράμματος της ε, Κροατίας ε, κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας για τους επόμενους μήνες και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ξεκινάμε με τους συντονιστές, ο κύριο Ντόρφμαν, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, σας καλωσορίζουμε θερμά. Κύριε Υπουργέ, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχω να προσθέσω πάρα πολλά σε αυτά που είπατε, γιατί με τα περισσότερα συμφωνώ. Κυρίως με αυτά που αναφέρατε για την κοινή γεωργική πολιτική. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο στο ότι τα κονδύλια πρέπει πράγματι να φτάνουν σε εκείνους που καθορίζουν ε, τη γεωργία Αναφέρομαι προφανώς στις ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ε, εκμεταλλεύσεις οι οποίες, ε, όπως σας είπα, είναι καθοριστικές για τη γεωργία αλλά και για το περιβάλλον. Σας παρακαλώ λοιπόν να μεριμνήσετε στο Συμβούλιο ε, ώστε να αναγνωριστεί το θέμα αυτό γιατί πολλές φορές εκφωνήθηκαν πανηγυρικοί αλλά όταν πρόκειτο για το ποιο τελικά θα είναι ο αποδέκτης, ο τελικός αποδέκτης των κονδυλίων εκεί τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Όλα αυτά βέβαια σχετίζονται και με την βιωσιμότητα. Εγώ εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, σήμερα είναι ε, βιώσιμες ή προσπαθούν να είναι βιώσιμες, γιατί οι ίδιοι οι γεωργοί δεν θέλουν να καταστρέψουν το έδαφος που καλλιεργούν ε, ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα. Εξορισμού οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις ε, είναι βιώσιμες, ενδιαφέρονται δηλαδή για την επιβίωσή τους, για την παράδοση της επιβίωσης στην επόμενη γενιά, γιατί μιλάμε ε, κατά κύριο λόγο για οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Ε, πολλές φορές ε, σήμερα ασκείται κριτική, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι όπως σας λέω σε γενικές γραμμές η διαχείριση είναι βιώσιμη. Όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις. Έχετε απόλυτα δίκιο. Ε, πρέπει να περάσει αυτός ο τεχνικός κονισμός το συντομότερο δυνατόν όσον αφορά τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, αυτή η στρατηγική θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τους επόμενους μήνες το agri-fish ε, θα πρέπει να παραμείνει κάτι σημαντικό, ουσιαστικό και εδώ στο Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι πολλοί προσπαθούν αυτό το θέμα να το αφαιρέσουν από τη γεωργία και να το περάσουν στην πολιτική υγεία, στην πολιτική διατροφής αλλά ξέρετε αν γίνει αυτό τελικά οι γεωργοί θα παραμείνουν απλοί θεατές. Γι' αυτό θεωρώ ότι agri-fish είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την βιώσιμη γεωργία. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπατε. Σα εύχομαι τα καλύτερα για του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά ε, καλώ ορίσατε, κυρία Μπουτσκοβιτ, ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Η Προεδρία τη Κροατία θα είναι πολύ σημαντική για τη Γεωργία. Αυτοί οι έξι μήνε θα ορίσουν επισήμως τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εύχομαι και τη θέση του Συμβουλίου. Ιδιαίτερα ε, όσον αφορά τις τρεις ε, νομοθετικές πράξεις ε, που τροποποιούν την κοινή κυρική πολιτική. Και εύχομαι πραγματικά να δημιουργηθούν οι καλύτερες προϋποθέσεις για να μπορέσουν και οι τριμερείς να φτάσουν σε αίσιο Εσείς μιλήσατε για το Πράσινο Σύμφωνο. Είμαστε υπέρ αυτής της μεγάλης που θέλησε να δώσει η Ursula von der Leyen και ολόκληρη η Κομισιόν. Πιστεύω πω η Γεωργία μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό, κρίσιμο ρόλο σε αυτή την πρόκληση του νέου ε, Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου. Αλλά για να το πράξουμε αυτό χρειαζόμαστε και γεωργική πολιτική η οποία να μένει σταθερά ε, αγκιστρωμένη στην Ευρώπη. Να μην υπάρχει κανένα κίνδυνος να μπορεί να επανεθνικοποιηθεί μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία έχει αποτελέσει ε, στις καλές και στις κακές μέρες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της ε, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Δεν θέλουμε λοιπόν να εθνικοποιηθεί ε, που να περιορίζει τις παρεμβάσεις ε, στα 27 κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν το τέλος της κοινή πολιτικής και γι' αυτό είναι πολύ ουσιαστικό το να διατηρήσουμε ένα κοινό όραμα και για να το καταφέρουμε αυτό, πιστεύω πως μία από τις μεγάλες καινοτομίες αυτής της πρότασης μεταρρύθμισης, το αυτή η δέσμη των πράσινων μέτρων θα πρέπει να αποφασιστεί και να, να οικοδομηθεί και να αποφασιστεί στις Βρυξέλλες. Και εντάξει, τα κράτη-μέλη θα έχουν μετά την ευθύνη να το εφαρμόσουν. Θα είναι ενδιαφέρουσα η, η, επαφή με την Κροατική Προεδρία και θα είναι πολύ σημαντική και για το ρόλο που θα παίξει το Κοινοβουλίο. Και για να τα καταφέρουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε και χρόνο αλλά χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τις συνθήκες ε, των γεωργών μας. Θα πρέπει αμέσως να πούμε στους γεωργούς μας ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα προχωρήσει και γι' αυτό χρειάζεται αυτή η μεταβατική, αυτός ο μεταβατικός κανονισμός. Συμφωνώ πως πρέπει να είναι ένας τεχνικής φύσης κανονισμός που θα εγκριθεί στα γρήγορα, αλλά όπως πάντα συμβαίνει με τις ε, κανονισμούς της συναπόφασης, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ε, να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν κάποιες μικρές ε, αλλαγές, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Καλή επιτυχία λοιπόν σας εύχομαι και είστε επανειδήν πολύ σύντομα. Πολύ ωραία να σας υπενθυμίσω ότι να κρατάμε λιγάκι το χρόνο που προβλέπετε για τον καθένα γιατί τελείως θα καταλήξουμε στο να χάσουμε τον έλεγχο. Να σας πω κάτι, επειδή ε, μία διερμηνέας αρρώστησε Σουηδικά ε, μπορείτε να μιλάτε, αλλά δεν θα μπορείτε να ακούτε Σουηδικά. Το λέω τώρα γιατί στην αρχή δεν μου το είχαν πει και δεν ήξερα κι εγώ να σας το πω. Ε, κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Θα ήθελα επίσης να σας συγχαρώ γιατί η Κροατία είχε πολύ καλή παρουσίαση στην, στα εγγένεια της Διεθνούς Πράσινης Εβδομάδας στο Βερολίνο. Όλοι οι Γερμανοί σας συμπάθησαν και ε, κατά την ε, τελευταία ε, συνάντηση που είχαμε μπορέσαμε να δούμε πώς ακριβώς είναι διαρθρωμένη η χώρα σας. Για μένα δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά. Αφενός σας ερωτώ, πιστεύετε ότι οι στόχοι ε, της Πράσινης Συμφωνίας πρέπει να ενταχθούν ε, στην κοινή γεωρική πολιτική. Γιατί ανησυχώ πάρα πολύ με την κοινή γεωρική πολιτική να περιμένουμε να ανακοινωθεί αυτή η περίφημη Πράσινη Συμφωνία. Ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω περαιτέρω ε, Και αυτό δεν θα βοηθήσει. Και μία άλλη ερώτηση. Το Συμβούλιο προτίθεται να προβεί σε ε, εκτίμηση του κόστους που θα επιβαρύνει τους ε, γεωργούς. Γιατί πάρα πολλοί περιμένουν πολλά από εμάς, την ευζοία των ζώων, τη βιωσιμότητα, την προστασία της βιοπικιλότητας. Όλα αυτά είναι προσδοκίες, αλλά ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει κόστος, τεράστιο κόστος που θα επιβαρύνει τη γεωργία. Και γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή ο τομέας λιανικής των τροφίμων δεν είναι πρόθυμος να πληρώνει περισσότερα στους γεωργούς για τα προϊόντα τους, ε, κάπου πρέπει να βρούμε μια ισορροπία, γιατί αλλιώς θα εξαφανιστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Κάπως πρέπει να ζουν και οι γεωργοί. Και αν δούμε λιγάκι τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ε, επιπρόσθετα κονδύλια, άρα δηλαδή εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για τις οικογενειακές, οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Εμένα με ενδιαφέρει στο πλαίσιο της ΚΑΠ να βρεθεί κάποια αξιοπιστία, να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις έτσι ώστε οι γεωργοί πράγματι να μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με μια βιώσιμη γεωργία που θα τους αρέσει πάρα πολύ. Ο κύριος Χόισλινγκ, κύριε Υπουργέ, ε, σας καλωσορίζουμε και εμείς θερμά. Ε, πράγματι, η εποχή που ζούμε είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί ε, και εσείς τελικά θα προτιμάσετε κάτι που θα τεθεί προς έγκριση ε, κατά τα τέλη του έτους. Υπάρχει εξή κατάσταση. Γίνονται διαπραγματεύσεις για μια κοινή γεωργική πολιτική. Αυτές ξεκίνησαν και με τον προηγούμενο επίτροπο. Όμως δεν είναι φιλόδοξη αυτή η πολιτική. Πάνω από 70% των κονδυλίων καταβάλλεται με βάση το εκτάριο και όχι την απόδοση. Αυτό όμω δεν ταιριάζει πια στην εποχή μα, γιατί μιλάμε για την Πράσινη Συμφωνία, για τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο και ο συνάδελφο κ. Μιλού το είπε αυτό. Αυτά κάπως συγκρούνται και τελικά δεν ξέρω ε, πώς ακριβώς μπορεί κανείς τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τους εντάξει σε μια φιλόδοξη γεωργική πολιτική γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο ε, σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα. Εσείς είπατε ότι δυστυχώς τελικά ε, δεν θα στηριχτούν οι οικογενειακές ε, γεωρικές εκμεταλλεύσεις. Αυτοί δεν θα αποφεληθούν από την κοινή γεωρική πολιτική. Αυτές οι εκμεταλλεύσεις σιγά σιγά εξαφανίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη έχουμε μια Ευρώπη όπου όλο και περισσότεροι ε, μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων υφαρπάζουν την γη των μικρών γεωργών και πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Εμείς ως πράσινοι λέμε ότι ναι, θέλουμε να καταβάλουμε κονδύλια, αλλά με ε, βασικό όρο την απόδοση. Εσείς αναφερθήκατε στη βιοπικιλότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβουργό είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για το θέμα αυτό. Γιατί το θέμα της ε, βιοπικιλότητας, παράλληλα με την κλιματική αλλαγή, είναι το καθοριστικό πρόβλημα, το ουσιαστικότερο πρόβλημα τη επόμενη δεκαετία. Και εκεί ε, καλείται να τοποθετηθεί και η γεωργία. Αναφερθήκατε στην μείωση των ζυζανιοκτώνων, φυτοφαρμάκων. Ε, εκεί πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Εγώ θα ήθελα να πείτε κάτι και για τη βιολογική, τις βιολογικές ε, καλλιέργειες. Γιατί αυτό τουλάχιστον είναι μια ευκαιρία για τις ε, μικρές επιχειρήσεις και για τη δική σας τη χώρα, για να υπάρξει πρόοδος. Και τέλος, δεν μιλήσαμε καθόλου για τη χρηματοδότηση. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ο δεύτερος πυλώνας ε, στην κοινή γεωρική πολιτική να είναι ο πυλώνας που θα χάσει τα περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστούμε. Συνάδελφος Ντάβιτ, παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το να μην αντιμετωπίζουμε τη γεωργία ως παράσιτο. Αλλά δυστυχώς ε, αυτό βλέπουμε τώρα. Ε, το ακούμε πολύ συχνά στα μέσα ενημέρωση ότι η γεωργία είναι κάτι που βλάπτει. Και αυτό όχι μόνο στη δική μου τη χώρα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Ακούμε επανειλημμένα ότι η γεωργία είναι εκείνη που βλάπτει το περιβάλλον. Ε, και τι κάνουμε εμείς ώστε να μην υπάρχει πια αυτή η άποψη, ώστε οι άνθρωποι να κατανοήσουν ότι και η Γεωργία έχει τα δικά της, τα σημαντικά καθήκοντα και ότι πρέπει να ασχολείται κανείς και με την παραγωγή των τροφίμων και να μην εξετάζει τη Γεωργία μόνο κάτω από το πρίσμα του περιβάλλοντος. Υπάρχουν ε, χώρες που έχουν διαφορετική δομή γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν είναι μόνο μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Τσεχία ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για μας μια μέση γεωρική εκμετάλλευση είναι της τάξης των 134 εκταρίων. Εσείς τι πιστεύετε, αυτό σημαίνει ότι είναι μικρή ή μεγάλη η γεωργική εκμετάλλευση, γιατί αυτές είναι οι εκμεταλλεύσεις δικές μας που συμμετέχουν καθοριστικά στην συνολική παραγωγή τροφίμων. Και μία ερώτηση, τι πιστεύετε εσείς για την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματο χάρη από Ηνωμένε Πολιτείες, Κίνα ή χώρες Μερκοσούρ ή ακόμα και Βιετνάμ, όπου παρά τις υποσχέσεις οι έλεγχοι δεν είναι αποτελεσματικοί, ε, δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές όπως αυτές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή εμείς περιμένουμε να εφαρμόσετε συγκεκριμένα προγράμματα που θα αποδείξουν ότι μπορείτε να ελέγξετε όλα τα προβλήματα που ετέθησαν σήμερα επιτάπητος. Ευχαριστώ κύριε Σκούσμιουκ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ να σας, να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω θερμότητα για την παρουσία σας στην Επιτροπή Γεωργίας. Και ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της κρατικής Προεδρίας. Και ιδιαίτερος ε, το γεγονός ότι τονίσατε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και στη χώρα που εκπροσωπώ, την Πολωνία, οι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει αποτελούν το μεγάλο τμήμα των γεωρικών εκμεταλλεύσεων και χαίρομαι που αναγνωρίζετε τη σημασία στήριξης αυτών των μικρών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, έχω τρεις ερωτήσεις για τις μεταβατικές αυτές διατάξεις, για τον κανονισμό των μεταβατικών διατάξεων για το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυτές οι μεταβατικές διατάξεις να ισχύουν μόνο για το 2021. Δεν θα κρίνεται σκόπιμο Αυτές οι μεταβατικές διατάξεις ε, λόγω της περιπλοκότητας της κοινή διορικής πολιτικής να έχουν διετή διάρκεια, δηλαδή να μην ισχύει μόνο για το 2021 αλλά και για το 2022. Δεν κρίνεται και εσείς σκόπιμο και απαραίτητο να παραταθούν για ακόμη ένα χρόνο. Επίσης, φάνηκε ότι είστε υπέρμαχος ε, της ε, ελαστικότητας, της ευελιξίας ε, της μεταφοράς κονδυλίων από τον πρώτο στο δεύτερο πυλώνα. Υπάρχει αυτό το ποσοστό το 25%. Δεν θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η διάταξη και στο μεταβατικό κανονισμό. Επίσης, θα χρειαστεί κάποια συμπλήρωση ίσως ε, μέσω των μεταβατικών διατάξεων και από τον Εθνικό Προϋπολογισμό και δεν ε, προβλέπεται κάτι τέτοιο ε, μέχρι στιγμής στους στις μεταβατικές διατάξεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να ισχύσει και για το 2021 και για το 2022 η δυνατότητα συμπλήρωση των κονδύλιων αυτών. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Um, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Εγώ προέρχομαι από τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και ασχολούμαι με την αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής αλλά και ιδιαίτερως ασχολούμαι με το να ταξιδεύω σε ολόκληρη την Ιρλανδία ε, ψάχνοντας ψήφους για συγκεκριμένους υποψηφίους στις εκλογές. Και κάτι ακόμα με το οποίο ασχολούμαι είναι ότι ανακαλύπτω πως πολλοί γεωργοί ε, αισθάνονται ανήσυχοι για το ότι θα χρειαστεί να προβούν σε μαζικές αλλαγές και θα πρέπει να συμβάλλουν προς την ε, ε, μείωση των κλιματικών αλλαγών ε, ενώ δεν θα πάρουν επιπλέον χρήματα για να το κάνουν αυτό. Αυτό που είναι βέβαιο και σίγουρο είναι ότι πρέπει κάτι τώρα να κάνουμε και επιγόντω για να μπορέσουμε να μετριώσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Γιατί να ακούσουμε του επιστήμονε, οι ίδιοι που μα λένε ότι υπάρχει η βαρύτητα, δείτε πώ πέφτει το τηλεφωνό μου, οι ίδιοι ακριβώ ε, επιστήμονε μου λένε πω το παιδί μου που είναι 5 ετών τώρα, εάν δεν δράσουμε γρήγορα, πιθανότατα θα πεθάνει από την πείνα όταν θα είναι 48 ετών που εγώ είμαι σήμερα. Άρα λοιπόν έχουμε να, θα έχουν να κάνουν τα παιδιά αυτά με χιλιάδες ανθρώπους που δεν θα έχουν που να ζήσουν και θα αναζητούν τόπο να ζήσουν και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φρικτό μέλλον εκτός αν κάνουμε κάτι τώρα. Ενώ ακούω λοιπόν τους γεωργούς και τους ανθρώπους που ανησυχούν αν θα πληρωθούν ε, ε, για το ότι θα κάνουν κάποιες αλλαγές. Ε, απ' την άλλη βλέπουμε ότι πρέπει να το κάνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε κάποια χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί έχουμε έτσι τις περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες πράγματι να κάνουμε κάτι αν το πράξουμε σωστά. Εσείς πιστεύετε πως θα υπάρξουν χρήματα για αυτά. Είναι καλύτερα η Ευρώπη να προχωρήσει στο δρόμο του να κόβει την πίτα με τέτοιο τρόπο ώστε περισσότερα να πηγαίνουν για να αγοράζονται βόμβες, όπλα και σφαίρες αντί να, να δαπανώνται για να έχουμε τρόφιμα και να αποφύγουμε τις κλιματικές αλλαγές από μια ουδέτερη χώρα όπως η Ιρλανδία, αυτό έχει περισσότερο νόημα. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Έληξε λοιπόν ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε πέντε λεπτά να απαντήσετε στα ερωτήματα που ετέθησαν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριοι συντονιστές ε, των πολιτικών ομάδων, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τις ερωτήσεις σας και για την υποστήριξη που δείξατε στην Κροατική Προεδρία. Έχουμε ένα πρόβλημα μικρό με την ε, γερμανική διερμηνία. Ακούω τα γαλλικά από το κανάλι της γερμανικής καμπίνας. Καλώ συνεχίστε κυρία Υπουργέ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους θερμότατα για την υποστήριξη που δείξατε στην Κρατική Προεδρία και για τις ερωτήσεις που υποβάλατε. Πολλές από τις ερωτήσεις σας, πολλές από τις αμφιβολίες σας τις αστερνίζομαι κι εγώ. Σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική και τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις, θα ήθελα να σας πω ξεκάθαρα και στα ράτα ότι η κρατική προεδρία θα προετοιμάσει το έδαφος για τις ε, διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο και θα αξιοποιήσει τις προσπάθειες των προηγούμενων προεδριών. Ελπίζουμε ε, να προχωρήσουν και οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν και οι διαπραγματεύσεις για τη γεωργία. Πάντως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες ώστε να καταλήξουμε σε συμφωνία στο Συμβούλιο για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τις μεταβατικές διατάξεις τώρα, αναμένω ότι ο κανονισμός για την ευελιξία θα υιοθετηθεί ήδη στο επόμενο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας που θα γίνει στις 27 Ιανουαρίου, σε λίγες μέρες δηλαδή και ελπίζουμε μέχρι ε, τα μέσα του 2020 να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις και τους ε, άλλους κανονισμούς και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να θετήσουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο γιατί θεωρούμε ύψιστη προτεραιότητα τη συνέχιση, την απρόσκοπτη συνέχιση της καταβολής των ενισχύσεων στους γεωργούς κατά το 2021. Σε ό,τι αφορά την παράταση που ζητήσατε των μεταβατικών διατάξεων. Μέχρι στιγμής αυτό που προβλέπετε είναι οι μεταβατικές διατάξεις να ισχύσουν το 2021. Πάντως είμαι βέβαιη ότι θα βρεθεί ο κατάλληλος ε, ταχύτατος μηχανισμός και για παράταση, αν παραστεί ανάγκη για τέτοια παράταση. Πάντως, ο στόχος μας είναι το συντομότερο δυνατό να υιοθετηθεί το μεταρρυθμιστικό πακέτο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ για να προσδιοριστεί και το θέμα της χρηματοδότησης και των μεταβατικών διατάξεων. Επίσης, στηρίζουμε τις φιλοδοξίες για το περιβάλλον και το κλίμα. Αλλά θα πρέπει αυτές οι φιλοδοξίες να συνοδεύονται με κατάλληλη χρηματοδότηση. Γιατί εμείς είμαστε Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας. Θέλουμε να στηρίξουμε τους γεωργούς, τους κοινοτρόφους και τον πληθυσμό της ε, των αγροτικών περιοχών και να διαφυλάξουμε την ανταγωνιστικότητα της γεωργικής παραγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις τρίτες χώρες. Σίγουρα θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να υιοθετήσουμε τον, και να υλοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό στόχο για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνεισφορά των γεωργών και, και με περικοπή του γεωργικού προπολογισμού. Είναι προφανέ ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθούν όλα αυτά αν περικόψουμε τον γεωργικό προπολογισμό. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, είχαμε ήδη στις 11 Δεκεμβρίου την παρουσίαση ε, της ε, Νέας Πράσινης Συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Εγώ θα αναφερθώ στις γεωρικές πτυχές αυτής της ευπρόσδεκτης ε, πρωτοβουλίας για τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Ε, πολύ σημαντική είναι η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Η Κρατική Προεδρία δεν θα αφιστεί προσπαθειών ώστε να διευκολύνει τις επικοδομητικές συζητήσεις στο Συμβούλιο και να προσδιορίσουμε τις σχέσεις της κοινή γεωρικής πολιτικής και της μελλοντικής ε, στρατηγικής από το χωράφι στο πιάτο. Θεωρούμε ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά όχι μόνο κατευθύνσεις. Δεν θα πρέπει η στρατηγική να είναι ένα γενικό έγγραφο. Θα πρέπει να προβλέπει συγκεκριμένες δραστηριότητες και να προσδιορίζει τα μελλοντικά μας βήματα, ώστε να υλοποιήσουμε το στόχο της ε, καλύτερης υγείας ανθρώπων, ζώων και φυτών και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Επίσης, θα πρέπει να περιορίσουμε τη σπατάλη των τροφίμων. Μέχρι στιγμής, δυστυχώς, δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη καταφέρει να περιορίσουν τη σημαντική σπατάλη των τροφίμων. Οπότε, λαμβάνουμε υπόψη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές. Θα ληφθεί αυτό υπόψη και στα εθνικά στρατηγικά σχέδια. Μέχρι στιγμής ε, εξετάζουμε τη, τα θέματα αυτά και περιμένουμε τις νομοθετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή γεωργική πολιτική. Συμφωνώ ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει κοινή. Αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα και ευελιξία. Και θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα και την ευχαίρεια στα κράτη-μέλη να προσδιορίσουν ε, κάποιους κανόνες ε, που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητές τους, εφόσον όμως εμείς θα καθορίσουμε το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες και την ηλικιακή ανανέωση, ε, είναι στόχος, υπάρχουν κάποια κίνητρα και δίνονται ενάυσματα, αλλά δεν αρκεί αυτή η κατάσταση. Θέλουμε να αυξηθεί το κονδύλιο για τους νέους αγρότες. Επίσης, ε, δεν συμφωνούμε με τη μείωση του, των κονδυλίων για τον δεύτερο πυλώνα, γιατί ο δεύτερος πυλώνας έχει συμβάλει τα μάλα στην ε, μεταμόρφωση της γεωργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ε, πρώτες απαντήσεις. Ε, θα περάσουμε και σε άλλες ερωτήσεις τώρα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε σε ένα λεπτό. Ποιος? Ο κύριος Ανδριού. Εδώ, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ για τη φιλόδοξη εισήγηση που μας κάνατε για να το... και ευχαριστώ επίσης που απαντήσατε στο ερώτημα που αφορά την μετάβαση. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιορισμοί που μας υποχρεώνουν να πράξουμε, να ενεργήσουμε και η μετάβαση όσο μας αφορά θα είναι μεγάλη, διότι ε, είμαστε σε μια κατάσταση, το είπατε και εσείς, όπου έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική, έχουμε το PDP και έχουμε και το πράσινο σύμφωνο. Και όλα μεταξύ τους είναι αλληλένδετα. Είναι σαν την κότα και το αυγό. Εφόσον όμως ζητάμε από τη Γεωργία να παίξει σημαντικό ρόλο και πολύ σημαντικό ρόλο στην Πράσινο Σύμφωνο, θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω μέσα. Άρα λοιπόν, για τη μετάβαση Μιλήσατε για ένα χρόνο που μπορεί να προσαρμοστεί όμως, ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά συμφωνείτε ότι η μετάβαση θα πρέπει να γίνει με νέους πόρους. Συνάδελφος Αφράν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία. Στη Γεωργία τα πράγματα είναι περίπλοκο περίπλοκα. Πάντοτε υπάρχουν πιο σκληρές συνθήκες. Οι γεωργοί μας ε, πρέπει να παράγουν καλύτερα, με πιο υγιεινό τρόπο, αλλά είναι όλο ένα και πιο δύσκολο. Και μια δυσκολία που πλήττει όλους στην Ευρώπη είναι ε, ο, δισταγμός, η απροθυμία των νέων να ασχοληθούν με τη γεωργία. Εμείς ε, περιμέναμε ότι θα γίνει μια μετάβαση προς μια νέα γενιά γεωργών. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Τι κάνει η Κροατία σε αυτό το τομέα. Υπάρχουν προγράμματα για να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ασχοληθούν με τη γεωργία. Κάνατε κάτι συγκεκριμένο και θα προτείνετε κάτι συγκεκριμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ κυρία Υπουργέ που ήρθατε μαζί μας ε, ε, για να ε, μα εκθέσετε τις προτεραιότητες με τις οποίες είμαστε σύμφωνοι. Μετά από μήνες συζήτηση στο Συμβούλιο για τι διαπραγματεύσει ε, τις δημοσιονομικές, νομίζω ότι εσεί ε, θα πρέπει τώρα να καταγράψετε μεγαλύτερη πρόοδο, όσο γίνεται μεγαλύτερη, όσον αφορά το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο η Φινλανδική Προεδρία είχε κάνει την επιλογή να αυξήσει τον προϋπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική σε σχέση με την ε, πρόταση της Κομισιόν, αλλά αυτή η αύξηση δεν αντιστάθμιζε την περικοπή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν ίσχυε παρά μόνο για το δεύτερο πυλώνα εις βάρος του πρώτου. Οπότε το ερώτημά μου είναι απλό ενώ το Πράσινο Σύμφωνο θα επιβάλλει νέους υποχρεώσεις στους γεωργούς μας, ενώ θέλουμε να έχουμε νέες φιλοδοξίες για τη γεωργία στην Ευρώπη, ποιες είναι οι δικές σας φιλοδοξίες πιο συγκεκριμένα για την κοινή γεωργική πολιτική. Μπόκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσίασή σας ε, και εγώ θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Συγκεκριμένα να ακούσω τη δική σας την άποψη για το περίφημο κάπινγκ. Ε, μιλήσατε για την υποστήριξη των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων και νομίζω ότι ένα βασικό στοιχείο είναι ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των χιλίων εκταρίων, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει κάτι, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να εξηγήσουμε ε, πώς ακριβώς ε, εκταμιεύονται τα κονδύλια. Πώς είναι δυνατόν τα κονδύλια να τα παίρνουν οι ολιγάρχες. Η απάντησή σας με ενδιαφέρει. Και τελικά τα χρήματα που λείπουν για την υγειορική εκμετάλλευση, ε, τι ακριβώς θα κάνουμε για αυτό το θέμα. Η δική σας η χώρα, αλλά και η δική μου η χώρα έρχονται αντιμέτωπες με αυτά τα προβλήματα. Η υπεθρός... Ε, καταλείπεται όλο και περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ κατά πόσον υπάρχουν ενδεχομένω κάποια προγράμματα για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Μήπως τελικά υπάρχουν κάποια κονδύλια στο Περιφερειακό Ταμείο έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα στην, ε, για τη γεωργία που να αφορούν ε, γεωργούς με δεξιότητες αλλά και ηλικιωμένους ανθρώπους. Ευχαριστώ κυρία Αγγιλέρα. Κύριε Υπουργέ, χθε σας είδαμε στην Ελία, σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, οι συνάδελφοι μίλησαν ε, για άλλα θέματα. Εγώ θα μιλήσω για την ανάγκη προσδιορισμού του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου χωρί περικοπέ τη κοινή γεωργική πολιτική. Χρειαζόμαστε απαραίτητα κονδύλια στην ΚΑΠ. Δεν θα πρέπει να στείλουμε εσφαλμένο μήνυμα στη γεωργία μας και την κτηνοτροφία μας. Δεν μπορούμε από τη μια να απαιτούμε περισσότερα από τους γεωργούς, να έχουμε περισσότερες περιβαλλοντικές και κλιματικές απαιτήσει και να τους δίνουμε λιγότερα κονδύλια. Αυτό θα ήταν πολύ λάθος, πολύ λάθος δρόμος. Οπότε θα πρέπει και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να αφήνει τον απαραίτητο χώρο και τα απαραίτητα κονδύλια στην κοινή γεωργική πολιτική. Με την αναθεώρηση της ΚΑΠ προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στη νέα πράσινη συμφωνία Πιστεύω ειλικρινά ότι ο μεταβατικός κανονισμός δεν αρκεί να έχει έτη διάρκεια. Θα είναι ρηξικέλευθη η αναθεώρηση της κοινή ζωρικής πολιτικής. Δεν μπορεί με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια σε ένα χρόνο να κάνουν τη μετάβαση στα κράτη-μέλη. Εγώ θα έλεγα ότι δύο χρόνια θα πρέπει να είναι η διάρκεια του μεταβατικού κανονισμού και όχι μόνο ένα. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Κατάινεν είναι η συγγήτρια για τη μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ στην Κροατική Προεδρία καλή επιτυχία. Το θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η Κροατική Προεδρία να προσπαθήσει πραγματικά να προάγει την κοινή γεωρική πολιτική τόσο όσον αφορά την μεταβατική περίοδο αλλά και την κανονική περίοδο. Ε, πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα γιατί οι γεωργοί χρειάζονται συνέχεια. Παραδείγματο χάρη, ο μεταβατικός κανονισμός ε, θα τεθεί σύντομα σε εφαρμογή και είναι αλήθεια ότι οι γεωργοί ε, χρειάζονται συγκεκριμένους κανόνες και είναι επίσης σημαντικό ε, η γεωργία να είναι βιώσιμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ερωτώ λοιπόν, εσείς τελικά πώς θα μεριμνήσετε έτσι ώστε τα κρατημέλη να αντιμετωπίζονται με ισότητα, με ίδιους όρους. Παραδείγματο χάρη, στην Φινλανδία ισχύουν τελείως διαφορετικοί όροι από ό,τι πολλές φορές στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συνάδελφος Αμάρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, Άκουσα πολύ, πολλές φιλοδοξίες και μεγάλη υποστήριξη προς τους γεωργούς και χάρηκα γι' αυτό και σας ε, συγχαίρω. Ελπίζω στη διάρκεια του εξαμήνου να μην χάσετε αυτή σας ε, την ε, ορμή. Και θα ήθελα εγώ να υπογραμμίσω πολλά από αυτά που υπόθηκαν, να μην δώσουμε δηλαδή ε, λάθος μηνύματα προς τους γεωργούς. Θα πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι όλοι μας υποστηρίζουμε τους γεωργούς ε, της Ευρώπης. Όμως εδώ, αν ύστερα στο Συμβούλιο ή στην Κομισιόν δεν συνοηθούν ε, σε σχέση με τη χρηματοδότηση, άρα το μήνυμα ήταν λάθος. Ναι, λέμε πολύ ωραία, ναι, αλλά μετά δεν δίνουμε τα χρήματα που χρειάζονται. Στη μεταβατική περίοδο η κυρία Υπουργό υποστηρίζει ή όχι ότι πρέπει να συνεχίζουμε να πληρώνουμε για το σημερινό μοντέλο ε, πριν να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ή όχι. Ευχαριστώ κύριο Ζροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ε, καταρχήν ε, να σας ευχηθώ τα καλύτερα για την Προεδρία. Να πω, αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι το πώς ακριβώς αντιμετωπίσετε την εξωτερική σύγκληση. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχει όμως και η κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δυστυχώς υπάρχει και ανταγωνισμός ε, και μέσα στην κοινή αγορά και γι' αυτό σας ρωτώ τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε στις χώρες της Βαλτικής καταβάλλονται πολύ λιγότερα κονδύλια από ό,τι σε υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο το 70% των κονδυλίων που καταβάλλονται σε άλλε χώρε. Η γεωργία σε εμά συρρυκνώνεται. Ε, Δυστυχώ υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην Ήπεθρο. Πια μπάκα, παρακαλώ. Madame la Ministre, je suis moi-même agricultrice. Κυρία Υπουργέ, εγώ η ίδια είμαι γεωργός στη Γουαδελούπη, σε ένα υπερπόδιο γαλλικό έδαφος. Εμείς φτιάχνουμε φρότα και λαχανικά. Ε, ε, σας ευχαριστώ που ήρθατε και έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Ε, σκέφτεστε να απλοποιήσετε το διοικητικό κομμάτι για τους μικρούς ε, τι θα κάνουμε απέναντι στο υπερφιλελεύθερο μοντέλο που μας, μας προτείνει ένα μοντέλο ε, υπερβιομηχανοποιημένο. Για μένα η γεωργία είναι ένας τομέας που έχει στόχο να θρέψει τους ε, πληθυσμούς και να δώσει ένα σωστό μισθό μια σωστή αμοιβή στους γεωργούς. Ποια είναι ε, το δικό σας όραμα για το μέλλον της γεωργίας και για την νέα κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ. Χάζεκάμπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Πριν από δύο καλοκαίρια πήγα σε ένα μικρό λιμάνι της Κροατίας ε, ένα από τα μικρά λιμάνια για τη μεταφορά ζώων στην Ευρώπη και είδα ένα νερό τάβρο που τον φόρταναν ε, σε πλοίο με γερανό και μάλιστα το έκαναν και ηλεκτροσόκ. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το μικρό λιμάνι της Ριέκα, αν ακούμε σωστά το όνομα. Ε, και τα ζώα, κύρια Υπουργέ, έχουν αισθήματα, νιώθουν άγχος, ε, ε, στρες, φόβο ε, όταν μεταφέρονται με τέτοιες συνθήκες. Επίσης, όταν ε, χωρίζουμε τα νεαρά ζώα, τα νεογνά από τις μητέρες τους. Νιώθουν μεγάλο φόβο και πολύ άγχος. Μιλάμε για καλή μεταχείριση των ζώων. Ερωτώ λοιπόν, τι θα κάνετε για το σκοπό αυτό στην Ευρώπη, για να εξασφαλίσουμε την ευζοία. Ο κύριος Μπιτσότο. E Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Ε, πρώτα απ' όλα σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τους επόμενους έξι μήνες που είναι καθοριστική σημασία για τη γεωργία μας. Ε, Κοιτάξτε, αν θέλουμε να ε, προσπίσουμε το περιβάλλον, πρέπει να επενδύσουμε στη γεωργία και όχι να αφαιρέσουμε κονδύλια από τη γεωργία. Γιατί το να υπερασπίζεται κανείς ε, ε, τους γεωργούς, αυτό σημαίνει ότι προστατεύει 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους, οι οποίοι πρέπει να να μπορούν να τρώνε καλά προϊόντα στις πατρίδες τους. το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πάρα πολλοί κατέβηκαν στους δρόμους στην Εμίλια Ρωμάνια ε, με τα εξής προβλήματα το πρόβλημα της ε, ασιατικής εισβολής ε, που έχει καταστρέψει πολλές γεωργίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν οι που σκοτώνουν τα ζώα. Κατόπιν υπάρχει το πρόβλημα των φρούτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την τιμή. Πολλοί δουλεύουν κάτω από την τελική αξία ε, και θα, αν συνεχίσουν θα καταστραφούν. Τα μεγάλα αρπακτικά, τα ε, σαρκοφάγα ε, και αυτά αποτελούν τεράστιο πρόβλημα για τη Γεωργία. Για το θέμα αυτό, τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε. Γιώργιλ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Είπατε τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν με τις, βάσει τις ιδιαιτερότητές τους πώς θα υλοποιήσουν ε, και ποιους στόχους θα υλοποιήσουν. Μα οι στόχοι προβλέπονται ήδη στη συνθήκη της Λισαβόνας. Μιλούμε για απαγόρευση των διακρίσεων, για ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ήδη είναι προκαθορισμένοι αυτοί οι στόχοι στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνετε κάποια μελέτη για το κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι της Λισαβόνας, ιδιαίτερα το άρθρο που μιλά για απαγόρευση των διακρίσεων και για ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Γιατί στο πακέτο που προτείνεται ε, και στο πακέτο για το Brexit, το θέμα της ε, σύγκλησης ε, φαίνεται ότι δεν υλοποιείται. Δεν είναι σωστή η η ενίσχυση που δίνεται στους γεωργούς και δεν ανταποκρίνεται στις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σε ευχηθώ καλή τύχη σε αυτό το εντατικό εξάμεινο που έχετε μπροστά σας στην Κροατική Προεδρία. Έχω δύο ερωτήσεις που έχετε περιλάβει και στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Η πρώτη αφορά τις νέες τεχνικές βελτίωσης, NBT. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Η κροτική Προεδρία πώς θα χειριστεί αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των νέων τεχνικών βελτίωσης. Δεύτερον, ε, τα, έξυπνα, τα έξυπνα χωριά στις αγροτικές περιοχές. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ε, ομάδας που έγινε την περασμένη εβδομάδα, Έγινε μια πρώτη συζήτηση. Εσείς τι ιδέες έχετε για να αναδείξετε και να προωθήσετε την πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα. Σας ευχαριστώ. Περιμένω να φορέσετε τα ακουστικά σας. Έχω μία ερώτηση για τη νέα πράσινη συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, στην Πράσινη Εβδομάδα του Βερολίνου, κατέβηκαν στους δρόμους χιλιάδες γεωργοί, διαμαρτυρώμενοι και εκφράζοντας αμφιβολίες τους για το νέο Πράσινο Σύμφωνο. Και στην Ρουμανία δεν έχουμε κατανόηση ακόμη το εύρος αυτής της νέας Πράσινης Συμφωνίας. Ποιοι είναι οι όροι που θα πρέπει να πληρούνται, τι υποχρεώσει θα έχουν οι γεωργοί, θα είναι επαρκή η χρηματοδότηση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στι επιδοτήσει και στι άμεσε ενισχύσει μεταξύ των κρατών μελών. Τι θα πούμε λοιπόν στου γεωργού μα, Οι γεωργοί αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ταυτόχρονα συνάπτουμε εμπορικέ συμφωνίε με χώρε ή με ομάδε χωρών όπω στην περίπτωση ε, της Μερκοσούρ που επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων από χώρες που δεν τηρούν τις ίδιες ε, με εμά υψηλέ προδιαγραφές και πρότυπα. Ευχαριστώ. Η κυρία Φρετζιόνοβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να φέρω ένα πρόβλημα το οποίο το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Οι γεωργοί φοβούνται πάρα πολύ ότι το κόστος θα εκτιναχθεί στα ύψη λόγω του πράσινη συμφωνίας και όλων αυτών των μέτρων για το περιβάλλον. Ε, Βεβαίω και θέλουν να έχουν καλή ποιότητα υδάτων, ε, θέλουν και βιώσιμη γεωργία, Κάπω όμως πρέπει και να τα βγάζουν πέρα. Εμείς στην Τσεχία έχουμε πάρα πολλέ μεγάλες ε, επιχειρήσει, αλλά εγώ θέλω να στηρίξω και τις μικρές γεωργικέ εκμεταλλεύσεις. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό ότι και εσεί το θίξατε το θέμα αυτό. Και νομίζω ότι τελικά είναι προς το συμφέρον μας να επιβιώσουν και οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις. Αλλά ε, δυστυχώς ε, οποτεδήποτε προκύπτουν προβλήματα, οι μικρές είναι εκείνες που θυσιάζονται, οι μεγάλες τα καταφέρνουν μια χαρά. Τελικά τι πρέπει να κάνουμε για να επιβιώσουν οι μικρές επιχειρήσεις. Τι είδου μέτρα προτίθεστε να εισάγετε έτσι ώστε να υποστηρίξετε τις μικρές επιχειρήσεις. Ο κύριος Ευχαριστώ και καλημέρα σας κυρία Υπουργέ. Για τους τρεις στόχους που αναφέρατε, οι δύο πρώτοι δεν είναι προβληματικοί, δηλαδή η απλούστευση που είναι απαραίτητη της ΚΑΠ και η επικουρικότητα που θα επιτρέψει στις χώρες να έχουν ένα με ευρύτερο περιθώριο λιγμών στα εθνικά στρατηγικά του σχέδια. Αλλά για την τρίτη σας προτεραιότητα, την αηφορία ή τη βιωσιμότητα, αυτή δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Πρώτη ερώτηση. Ποια θα είναι η σχέση αυτού του στόχου της αηφορίας της γεωργίας με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ε, το ίδιο, τους ίδιους στόχους αυτά τα δύο προγράμματα ή το ίδιο θεματολόγιο. Ε, γιατί η ΚΑΠ έχει προχωρήσει αρκετά, ενώ η Νέα Πράσινη Συμφωνία βρίσκεται στα Σπάργανα. Πώς θα βοηθήσετε τους γεωργούς που ιδιαίτερα στην Γαλλία ε, θεωρούνται υπεύθυνοι για την... Ε, επιδείνωση της κατάστασης στο περιβάλλον. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στην αρχή είχε ενθαρρύνει τη μαζική χρήση των φυτοφαρμάκων, τώρα θέλει να τα μειώσει σταδιακά. Επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ των συμφωνιών ελεύθερων ανταλλαγών που θα επιτρέψει δυστυχώς εισαγόμενα προϊόντα που δεν τηρούν του κανόνες μας να εισαχθούν στη Γαλλία. Ε, κυρία Λινό. Äh, Καλημέρα σας ε, κύριε Υπουργέ, σας ε, καλωσορίζουμε στο Κοινοβούλιο. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής, ότι ε, πριν από λίγο καιρό επιστήμονες μας παρουσίασαν μία μελέτη που αφορά στις άμεσες ενισχύσεις, ε, πώς αυτές επηρεάζουν την ύπεθρο, τους ανθρώπους. Μας απέδειξαν ότι πρόκειται για στρέβλωση του ανταγωνισμού, ότι ε, πράγματι ε, σε πρώτη φάση υπάρχει μια υποστήριξη προς τις μικρές εκμεταλλεύσεις, αλλά τελικά μακροπρόθεσμα δημιουργείται πρόβλημα λόγω στρέβλωσης ανταγωνισμού. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ερωτήσω, στην Κροατία υπάρχουν εξαιρέσεις για να γίνουν γίνουν κάποιες ε, μεταφορές από τον δεύτερο πυλώνα στον πρώτο πυλώνα. Ε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί υπάρχουν ε, πάρα, πολλές, πάρα πολλά αιτήματα στον δεύτερο πυλώνα. Εσεί τώρα μπορείτε να είστε ένα πρότυπο για το πώ μπορεί να στηριχτεί η Γεωργία η και ρωτώ, έχετε προγράμματα που να στηρίζουν το δεύτερο πυλώνα στην Κροατία. Και το δεύτερο σκέλος ερώτησή μου είναι ότι βλέπουμε και θέλουμε το μέλλον να είναι βιώσιμο. Ποια είναι η άποψή σας για τη Μερκοσούρ και για τα δικαιώματα ε, ανταγωνισμού, για τον ίσο ανταγωνισμό. Όλοι θέλουμε να μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά αν πραγματικά το θέλουμε όλοι, τότε δεν θα πρέπει να καταλάβουμε ενισχύσεις με βάση την έκταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, ε, για το ότι δείχνετε να θέλετε να στηρίξετε τους Ευρωπαίους γεωργούς. Καταρχήν θέλω να πω, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σημαίνει, και αυτό πρέπει να το καθιστούμε σαφές, ότι η γεωργία είναι ο μόνος τομέας ο οποίος παράγει οξυγόνο, αλλά και δεσμεύει και διοξίδιο του άνθρακα. Κανένα άλλο δεν το κάνει αυτό. Δεύτερον, ε, μπορούμε να παρατηθούμε πολλά στη ζωή αυτή, αλλά δεν μπορούμε να παρατηθούμε από το φαγητό. Ε, και δυστυχώ αυτό πολλοί το ξεχνάνε. Ε, τρίτον, εσείς μιλήσατε για τον τετραγωνισμό του κύκλου. Έχουμε όλο και περισσότερα καθήκοντα, περισσότερους όρους και προποθέσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται όλο και λιγότερα χρήματα. Ε, και εγώ ε, θα κάνω το εξή ρητορικό ερώτημα. Τελικά, αν όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ας υποθέσουμε ότι τις μετατρέπουμε σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις, τότε τι θα γίνει. Θα υπάρχουν περισσότερα χρήματα, τότε θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ο συνάδελφος κύριος Γιάρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ως εισηγητής της κοινή γεωργικής πολιτικής χαίρομαι που θα συνεργαστούμε. Και κάποιες μικρές ερωτήσεις. Κατάλαβα καλά ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου ε, θα έχουμε κοινή άποψη του ε, Συμβουλίου για την κοινή γεωρική πολιτική. Το είπατε, το κατάλαβα καλά. Δεύτερον, μέχρι τις 30 Ιουνίου ε, θα έχουμε δημοσιονομικές προοπτικές, θα έχουμε προϋπολογισμό. Εσείς, αν κατάλαβα καλά, λέτε μάλλον όχι. Το τρίτο μου ερώτημα όσον αφορά την Πράσινη Συμφωνία. Εσείς τι πιστεύετε, την Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να τον εντάξουμε στο δικό μας τον ή θα υπάρξουν άλλα έκτακτα κονδύλια άλλη ερώτηση. Ενισχύσεις με βάση την έκταση. Ε, το έχουμε στήσει πολλές φορές. Ε, δεν βρήκαμε κάτι καλύτερο. Επανήλθαμε σε αυτή την μορφή ενισχύσεων και γιατί θέλουν πολλοί ε, στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις να καταργήσουν τις ενισχύσεις με βάση την έκταση. Μετά, τη γεωργία πιστεύετε θα πρέπει και στη γεωργία να ισχύει το σύστημα αυτό της ανταλλαγής εκπομπών. Συνάδελφος Φλάτσεκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την ε, διεξοδική παρουσίαση των προτεραιοτήτων της κρατικής προεδρίας που είναι και πολύ φιλόδοξες. Εγώ είμαι από την Τσεχία και έχουμε κάποιον στο Συμβούλιο που δείχνει κατανόηση στα κράτη-μέλη λόγω της διαφορετικής ιστορίας τους, αλλά και λόγω της διαφορετικής διάρθρωσης της γεωργίας τους. Έχετε ένα πολύ υπεύθυνο ρόλο γιατί αναλαμβάνετε την Προεδρία σε πολύ κρίσιμους μήνες ε, για τις φάσεις των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα πριν ε, καταφέρετε το χτύπημα, θα ήθελα να διαρωτηθείτε θα θέλουμε μια πιο δίκαιη ΚΑΠ και αν μετά την ε, διεκπαιρέωση της κρατικής προεδρίας. Η απάντηση είναι θετική, αν δηλαδή έχουμε καταλήξει σε μια δικαιότερη ΚΑΠ θα μπορείτε να είστε υπερήφανοι. Και όταν εννοώ δίκαιη ΚΑΠ, ενώ επιβραβεύουμε αρκετά τους ε, γεωργούς ε, για όλες τις νέες απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουμε. Επιβάλλουμε δίκαιους στόχους για τους γεωργούς ή μήπως περικόπτουμε τα κονδύλια και του στερούμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν του όρου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Σίντσιτ. Σα ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε για προτεραιότητα στην ενίσχυση του προπολογισμού της ΚΑΠ και προτεραιότητα στους μικρούς ε, γεωργικούς, ε, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. όμως την εμπειρία της Κροατίας και το πώς λειτουργεί η γεωργία, διαπιστώνω ότι αυτή η υποστήριξη στις μικρές ε, καλλιέργειες μόνο στη θεωρία υπάρχει. Ε, είναι μόνο ρητορική. Οι μικροί καλλιεργητές παίρνουν το 1 τρίτο μόνο των ενισχύσεων. Βλέπετε τη διαφορά. Επίσης, ε, δεν μπορούμε ε, ε, να δίνουμε 2 τρίτα των ενισχύσεων στις μεγάλες ενισχύσεις, ενώ το 97% των εκμεταλλεύσεων είναι μικρές εκμεταλλεύσεις. Ε, 240 ε, εκατομμύρια πήραν 70 ε, μικροί, ενώ τα διπλάσια πήραν ε, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις. Ένα τεράστιο ποσό πήγε σε λίγους παραγωγούς και ένα πολύ μικρό ποσοστό στους πολλούς παραγωγούς. Επίσης, λάβαμε πολύ λιγότερα από ό,τι έχουμε πληρώσει. Πληρώσαμε 3 δις και πήραμε μόνο 1,1 δις. Θα πρέπει αυτό να το λάβετε υπόψη στις προτάσει για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ, να εξασφαλίσετε ισορροπία μεταξύ των μεγάλων και μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν έχετε καταφέρει όμως δυστυχώς να αποκαταστήσετε ούτε μέσα στην Κροατία. Σας ευχαριστώ. Σμιτ Μπάουερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις φιλόδοξες απόψει σας ε, και ε, για τι υποσχέσει που μας δώσατε. Εδώ είμαι, κύριε Υπουργέ, από την Αυστρία έρχομαι, ξαναρχίζω. Ευχαριστούμε πολύ για τους φιλόδοξους ε, στόχους σας. Ε, ως Αυστριακή ε, χαίρομαι για τη συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας στηρίξω όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις. Και να στρέφομαι και προς τους συναδέλφους. Πρέπει να καταλήξουμε σύντομα και για όνομα του Θεού να μην φτάσουμε και πάλι σε μία μικρή μεταρρύθμιση. Ένα πράγμα, επ' αυτού συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, ότι θέλουμε να ασχοληθούμε και να ενισχύσουμε περισσότερο τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αυτές οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται ασφάλεια. Να μην καταλήξουμε σε μία μίνι μεταρρύθμιση, να συζητήσουμε, να τα βρούμε για την κοινή γεωρική πολιτική και τώρα πρέπει να αρχίσει να ρέει το χρήμα. Ε, τώρα το θέμα των περικοπών στο δεύτερο πυλώνα, αυτό για μας θα ήταν καταστροφή. Εμείς έχουμε επιλέξει ένα πολύ καλό σύστημα. Ε, σε εμά ε, στην Αυστρία το 1 τρίτο είναι άμεσε ενισχύσει και τα 2 τρίτα διοχετεύονται στην ανάπτυξη. Αν λοιπόν θέλουμε να ε, διατηρήσουμε τις γεωργικέ εκμεταλλεύσεις, τότε δεν πρέπει επουδενή να καταλήξουμε σε αυτές τις τεράστιες περικοπές. Άρκοβιτς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση και βλέπω ότι είναι και πάρα πολλοί στόχοι, ενώ τα κονδύλια δεν επαρκούν. Έχουμε και τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Θα ήθελα ε, να επικεντρωθώ στην πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά. Ξέρω ότι η Κροατία κάνει αρκετές προσπάθειες και διασυνοριακά εφαρμόζει αυτό το σχέδιο για τα έξυπνα χωριά. Τι γνώμη έχετε και τι εμπειρία έχετε αποκομίσει από την εφαρμογή αυτού του σχεδίου στο... μέχρι στιγμής. Ο κύριος Γκερέρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια πολύ σύντομη και άμεση ερώτηση σε σχέση με τις έρευνες που έγιναν από το New York Times και που συνδέουν την, ε, τα χρήματα της γεωργικής πολιτικής που δόθηκαν σε πολλές χώρες ε, με την ανάπτυξη ε, δικτατορικών τάσεων και των ολιγαρχών σε ορισμένες χώρες. Τι έχετε να πείτε για αυτά όλα. Εδώ μιλάμε για την κοινή γεωργική πολιτική η οποία πρέπει να ενισχύει μόνο και αποκλειστικά τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω κυρία Υπουργέ για τους επόμενους έξι μήνες εύχομαι καλή επιτυχία και θέλω να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε ένα από τα δράματα που θα πρέπει να μας ε, κάνουν να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ε, στην ε, στα πλαστά διατροφικά προϊόντα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πλήττει τους γεωργούς μας, ε, την τεχνογνωσία τους, ε, την εμπειρία τους και μπορεί να είναι επικίνδυνο και για την υγεία των πολιτών. Μπορείτε να μας δώσετε κατευθύνσεις για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ε, πολλές ερωτήσεις ε, και τώρα θα περάσουμε στις ε, απαντήσεις. Θα έλεγα λοιπόν να σας διαθέσουμε περίπου 10 λεπτά. 10 λεπτά, κυρία Υπουργέ, να προσπαθήσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Poštovane zastupnice i zastupnici, hvala na svim vašim pitanjima i korisnim sugestijama. Bilo ih je mnogo, doista ću nastojati barem ukratko. ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Για τις... Ε, θα μιλήσουμε για τον κανονισμό, για τη μεταβατική περίοδο ε, και βεβαίως Όλα αυτά γίνονται με βάση των προηγούμενων διαθέσιμων ε, για νέα χρήματα. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο όμως για να μπορέσουμε να εισάγουμε μία πηγή ε, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. Συμφωνώ και καταλαβαίνω τις αμφιβολίες σας και ξέρω ότι ίσως ένας χρόνος είναι πολύ περιορισμένο διάστημα αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα. Προς το παρόν, προτεραιότητά μας είναι να καθορίσουμε τους κανόνες. Ίσως χρειαστεί παράταση, αλλά θα το δούμε αργότερα. Το βασικό είναι να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία για τους μεταβατικούς ε, κανόνες μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας όλα τα θέματα, περιμένουμε ε, και τις συμφωνίες και για το ΠΔΠ. Πάντως, στόχος μας είναι να καθοριστεί το πλαίσιο, τουλάχιστον. Σε ό,τι αφορά τη σχέση της κοινή γεωργικής πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, σίγουρα η ΚΑΠ ε, είναι σε προωθημένη φάση και εντάσσεται και στην... Ε, ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τη Νέα Πράσινη Συμφωνία, αλλά οι γεωργοί μας ήδη εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζουν τη δημοσιότητα. Και ένα τμήμα της ανακοίνωσης για την ε, νέα πράσινη συμφωνία ήδη αποτελεί τμήμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εμείς θα ε, επικεντρωθούμε στη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Θέλουμε να συγκεκριμενοποιηθεί, να συνοδευτεί από συγκεκριμένες δράσεις και δραστηριότητες, να περιλαμβάνει μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων, την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της και την αναζήτηση εναλλακτικών ε, φυσικών ε, τρόπων καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών. Επίση θέλουμε να καταπολεμήσουμε την σπατάλη των τροφίμων και να δώσουμε έμφαση στην καλή μεταχείριση των ζώων. Η ευζοή είναι πολύ σημαντικό θέμα, το είπα και στην αρχική μου ομιλία και συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα ε, περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανταποκριθεί στην έκκληση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καλή μεταχείριση των ζώων και να υποβάλει τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις, αλλά και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις, γιατί οι διατάξεις υπάρχουν για την καλή μεταχείριση των ζώων από το 2011. Θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εξασφαλίζονται σωστοί έλεγχοι. Πάντως, στι 27 Ιανουαρίου στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλίας, το θέμα τη ευζοή και τη καλή μεταχείριση των ζώων περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξωτερική σύγκληση και το κάπινγκ, τα ανώτατα όρια. Είχαμε δύο ερωτήσεις για την εξωτερική σύγκληση και μία ερώτηση για το κάπινγκ, τα, τις οροφές και τα δύο θέματα βρίσκονται στο κουτί των διαπραγματεύσεων. Αυτό που μπορούμε να πούμε ως κρατική Προεδρία είναι ότι όντως υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και για τα δύο θέματα, και για το κάπινγκ και για την εξωτερική σύγκληση. Εμείς ε, θα λειτουργήσουμε ως διαμεσολαβητές για να υπάρξει μια σύγκληση των απόψεων και το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο φυσικά και η συζητήσει εκεί θα επηρεάσουν το διαπραγματευτικό περιεχόμενο και αυτών των προτάσεων. Η πρωτοβουλία για τα έξυπνα χωριά είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ο δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ προβλέπει την βελτίωση των συνθηκών προκειμένου να παραμείνει ο πληθυσμός στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Και αφορούσε περισσότερο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στην Ήπεθρο. Εμείς στηρίζουμε τέτοια μέτρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εφαρμόσαμε και στην πατρίδα μου την Κροατία. Και σίγουρα δεν αρκεί να έχουμε μόνο καλύτερες ε, υποδομές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε και άλλες ε, έννοιες για να υλοποιήσουμε τα έξυπνα χωριά. Και θεωρώ ότι με μια τέτοια πρωτοβουλία θα υλοποιήσουμε το στόχο μας να προσελκύσουμε κόσμο στην Ήπεθρο και να κρατήσουμε τον πληθυσμό στην Ήπεθρο και φυσικά ε, να προσελκύσουμε και νέους στην Ήπεθρο. Όλες οι εκμεταλλεύσεις είναι απαραίτητες στην Ευρωπαϊκή Γεωργία, και οι μικρές και οι μεσές και οι μεγάλες. Όλες χρειάζονται στη γεωργία και στην οικονομία. Θα πρέπει ε, να στηρίξουμε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και στην οικονομία και στη γεωργία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να στηρίξουμε τις μικρές καλλιέργειες, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, γιατί έτσι θα κρατήσουμε τον ε, αγροτικό πληθυσμό στην Ήπεθρο. Και φυσικά θα επιδιώξουμε και μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Αυτές τις συζητήσεις θα προωθήσουμε στο Συμβούλιο και γι' αυτό η Κροατική Προεδρία θα οργανώσει και μια ειδική διάσκεψη με θέμα το παρόν και το μέλλον των οικογενειακών και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Επίσης, μιλήσατε για την αξιοποίηση των περιφερειακών κονδυλίων είχα ασχοληθεί με την εφαρμογή και τον έλεγχο των διασυνοριακών προγραμμάτων. Αυτές ήταν οι πρώτες εμπειρίες εργασιακές που είχα για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ήδη υπάρχει δυνατότητα, λόγω των πολλών διασυνοριακών προγραμμάτων, να απορροφηθούν και κάποια περιφερειακά κονδύλια. Και θα μπορούσαμε στα προγράμματα αυτά να συμπεριλάβουμε και κάποια στρατηγικά προγράμματα που εύκολα θα συμβάλλουν στην αγροτική ανάπτυξη. Εγώ από την προηγούμενη εμπειρία που είχα για τη διαχείριση των διασυνοριακών προγραμμάτων και για την, με τη νέα γενιά των διμερών προγραμμάτων με τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και άλλες χώρες, διαπιστώνω ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα και ανάλογα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουμε μπορούμε να απορροφήσουμε συμπληρωματικά κονδύλια που θα υλοποιούν τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής. Τέθηκε μία ερώτηση και για τις νέες τεχνικές βελτίωσης. Φαντάζομαι να φέρεστε και την σχετική νομολογία του 10 του 2011. Με την απόφαση του ΔΕΚ δημιουργούνται πολλές ευβολίες και ανοίγουν πολλά πρακτικά θέματα θα πρέπει με βάση την ομολογία αυτή να κανονίσουμε και τη μελλοντική μας ε, νομοθεσία. Ε, πάντως, ε, το Συμβούλιο ζήτησε στα τέλη του 2019 μελέτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, φάση των νέων, για τη φάση στην οποία βρίσκονται οι νέες τεχνικές βελτίωσεις υπό το φως και τη σχετικής νομολογίας του ΔΕΚ. Περιμένουμε λοιπόν αυτή τη μελέτη, αυτή την έρευνα που ζήτησε το Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλογα με τα πορίσματα που θα λάβουμε από την μελέτη αυτή θα ε, συνεχίσουμε τη συζητήση στο Συμβούλιο. Τέθηκαν και τρεις ειδικέ ερωτήσεις για την Κροατία. Αναφερθήκατε σε μία υπόθεση πριν από μία τριετία, ε, μία περίπτωση παραβίασης ε, των αρχών καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά στο μεταξύ λύθηκε το θέμα, έγιναν πιο αυστηροί έλεγχοι στην Κροατία και δεν επαναλήθηκε αυτό το φαινόμενο κακής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά. Επαναλαμβάνω, από τότε που εφαρμόσουμε την κοινή γεωρική πολιτική, ο αριθμός των γεωργών αυξήθηκε κατά 2.000 και μάλιστα έχουμε και πολλούς ε, ε, νέους γεωργούς. Το 13,1% των γεωργών μας είναι νεαροί αγρότες. Έχουμε μεγάλη βελτίωση και είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν θα επαναπαυθούμε σε αυτή την επιτυχία. Θέλουμε να προσαρκίσουμε ακόμη περισσότερους νέους για να εξασφαλίσουμε και την ηλικιακή ανανέωση. Υπάρχει μάλιστα ειδικό κονδύλιο για τους νεαρούς αγρότες και στις άμεσες ενισχύσεις, αλλά και στο Γενικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. 1.500 ε, προγράμματα έχουμε χρηματοδοτήσει ε, ύψους 520 εκατομμυρίων κούνων. Δεν ξέρω πόσο είναι σε ευρώ. Τέθηκε και μία τρίτη ερώτηση για την Κροατία, τη διαφορά των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Έχουμε συγκεκριμένο κονδύλιο για τις άμεσες ενισχύσεις και παρόλο που ήταν θέμα εθνικό, θα σας απαντήσω συγκεκριμένη κυβέρνηση προσπάθησε να δώσει ε, έμφαση και μεγαλύτερη προτεραιότητα στις μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, ώστε να καρπώνονται ένα μεγαλύτερο τμήμα των άμεσων ενισχύσεων από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση και επιτρέπουμε όλος, όλο, σε όλο και περισσότερους μικρούς καλλιεργητές να υποφελούνται από προγράμματα και κονδύλια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε άλλωστε και ξεχωριστούς διαγωνισμούς στα προγράμματα μεταξύ μικρών και μεγάλων καλλιεργητών. Και το μέτρο 4 ειδικά για τις επενδύσεις δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. 60% των κονδυλίων πήγε στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις και 40% του κονδυλίου πήγε στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να καθοδηγηθούμε όχι μόνο από το μέγεθος εκμετάλλευσης, αλλά και από το μέγεθος της παραγωγής και το μερίδιο της αγοράς. Πάντως θέλουμε μια πιο δίκαιη κατανομή των κονδυλίων. Η Κροτή βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία του phasing in. Και το ποσό που αναφέρει των τριών δισεκατομμυρίων είναι το ανώτατο ποσοστό. Ε, μέχρι στιγμής ε, ε, είχαμε δυνατότητα και όχι υποχρέωση. Και επίσης τηρήσαμε τις διατάξεις και για τη συμπλήρωση με εθνικά κονδύλια στο μέτρο του δυνατού και, και το 70% του, του συνολικού κονδυλίου το έχουμε απορροφήσει και νομίζω ότι είναι αρκετά ικανοποιητικό αυτό το ποσοστό και για το 2020 περιμένουμε να έχουμε εκταημίευση του συνόλου του εθνικού κονδυλίου, το 100% δηλαδή, που είναι μεγάλη πρόοδο σχέση με το 70% απορρόφηση που είχαμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι απλό να απαντήσει κανείς σε 25 ερωτήσεις μέσα σε 10 λεπτά ε, και στις ε, ερωτήσεις που ετέθησαν κρύπτονταν και άλλες μικροερωτήσεις. Έκανα και ένα μικρό λάθος. Την ξέχασα τη συνάδελφο Τόμασιτς παρότι την είχα ε, στο κατάλογο μου. Κύριε Τόμασιτς, γι' αυτό το λόγο, σας δίνω το λόγο για να κάνετε μια ερώτηση για ένα περίπου λεπτό. Κυρία Τόμασιτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε και καλή τύχη στην Κροατική Προεδρία. Άκουσα τις απαντήσεις ε, στις ερωτήσεις. Θα ήθελα μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. Σίγουρα ανοίγουν και ξεκινούν πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις, αλλά και πολλές αντίστοιχα κλείνουν και βάζουν λουκέτο. Πώς προβλέπετε να στηρίξετε τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και τι δράσεις θα αναλάβετε ώστε να προσελκύσετε νεαρούς αγρότες, να εξασφαλίσετε τον εξυγχρονισμό της γεωργίας και να ενισχύσετε ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, πριν λοιπόν ε, ε, δώσω το λόγο ε, και πριν κάνει και την τελική της δήλωση, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να δώσω ε, σύντομα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν δεν θέλετε, καλά. Αφού δεν θέλετε, πολύ καλά. Ε, τότε να δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό για να μας απαντήσει και για να κάνει και την τελική της δήλωση. Σας ευχαριστώ, κύριε Τόμασιτς. Εκτός ότι θα οργανώσουμε μια διεθνή διάσκεψη για το μέλλον των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, θα προσπαθήσουμε και στο Συμβούλιο να προωθήσουμε την υποστήριξη το, της απλούστευσης τον κανόνων της ΚΑΠ για τις μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, η απλούστευση για τους μικρούς καλλιεργητές. Θέλουμε να απλουστεύσουμε τη γραφειοκρατία και τη διαδικασία και να βελτιώσουμε την πρόσβαση των μικρών καλλιεργητών στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να απολαμβάνουν τους καρπούς της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και μια και απάντησα προηγουμένως στις ε, προηγούμενες ερωτήσεις, ε, σας Επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, η γεωργία δεν είναι πρόβλημα, είναι τμήμα της λύσης. Θα πρέπει λοιπόν να, να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη γεωργία, αν την αντιλαμβανόμαστε ως κίνδυνο ή πρόβλημα. Δύσκολο είναι να βρει κανείς άλλο, τομέα που να είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο όπως είναι η γεωργία και η Αλία. Και νομίζω ότι η γεωργία ε, είναι ο τομέας που προστατεύει τον άνθρωπο, το περιβάλλον, την υγεία, τους φυσικούς πόρους. Και άλλωστε η γεωργία ήταν ανέκαθεν φορής καινοτομίας. Λάθος πιστεύουν μερικοί ότι η γεωργία είναι αντιδραστική και ότι δεν υπάρχει καινοτομία στη γεωργία. Άλλωστε δεν υπάρχει πιο ευγενής μορφή οικονομικής δραστηριότητας από τη γεωργία και την αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Υπουργέ ε, για την παρουσία σας, ε, για τις ε, διεξοδικές απαντήσεις που δώσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε τους επόμενους έξι μήνες. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και σημαντικά και χαίρομαι πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.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 So, dear, dear colleagues, please take your seats again. We will continue the meeting and we... Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση και να φτάσουμε και στις ψηφοφορίες. Μάλλον να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Good morning.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ε, λιγάκι έχουμε καθυστερήσει. Πάμε τώρα στο σημείο υπερθμών 5 Τη ημερήσιας διάταξης σε τρεις ε, ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με το σημείο υπερθμών 5. Ε, πρόκειται για τη σύναψη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομική ενέργεια. Μήπως η συγγήτρια επιθυμεί να λάβει το λόγο πριν από την ψηφοφορία, συνάδελφος κύριε Μακίνης. Όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ως εκ τούτου μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις ε, κάρτες σας, τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ε, και η τελική ψηφοφορία, όπως πάντα, θα γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν παρακαλώ. Ich äh, schließe die Abstimmung. Έκλεισε η ψηφοφορία. Ist, ist angenommen. Εγκρίνεται. Δεκτό ε, με 43 ψήφους. Συγχαρητήρια. Περνάμε τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ξέρω, όπω είπατε, συγχαρητήρια, αλλά με πολύ βαριά καρδιά στηρίζουμε αυτή την έκθεση και με πολύ βαριά καρδιά το συντάξαμε κιόλα αυτό το ψήφισμα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία του να αποχωρήσει ένα μεγάλο κράτος μέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και να, την εκφράσω την εκτίμησή μου στου συναδέλφου από την Βρετανία που ήταν πολλά χρόνια εδώ σε αυτή την Επιτροπή, πολλοί εξ αυτών φίλοι, καλοί συνάδελφοι και ξέρω πω είναι δύσκολη στιγμή για πολλού εξ αυτών. Vielen Dank. Πάμε τώρα στην ε, γνωμοδότησή μας για, τον, για την πολιτική ανταγωνισμού. Πολιτική ανταγωνισμού λοιπόν. Η έκθεση 2019. Η συγγήτρια η κυρία Καρβαλές επιθυμεί να λάβει το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα μικρό σχόλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ε, καλή του συνεργασία. Ήταν πολύ παραγωγικό και καρποφόρο το έργο μας και θα ήθελα να εξάρω το πνεύμα συνεργασίας που επέδειξαν ε, όλοι οι συνάδελφοι και να ευχαριστήσω και τους βοηθούς μου. Καταφέραμε να συντάξουμε γνωμοδότηση που εστιάζεται στις πιο σημαντικές αρχές και παρόλα αυτά καταφέραμε να συντάξουμε μια στέναρη άρτια γνωμοδότηση κρατώντας ε, όμως μια συνοπτική διατύπωση επικεντρωμένη σε λίγες και σημαντικές αρχές. Επίσης δεχτήκαμε και μια προφορική τροπολογία ε, και έτσι περιλάβαμε τις τροπολογίες 87 και 90 με τη συνοπτική προφορική τροπολογία. Η προφορική τροπολογία λοιπόν περιλαμβάνεται και αυτή στην έκθεση και ήταν ανέκαθεν πρόθεσή μας να κρατήσουμε μια ευσύνοπτη γνωμοδότηση που θα επικεντρώνεται στις ε, βασικές αρχές που διαμορφώνουν μια σημαντική, στεναρή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια για τη δουλειά τη. Προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία, αλλά πρώτα δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Λεμπρετόν. Πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου για τι τροπολογίε 28 και 67. Αναφέρεται ότι καλύπτονται από την συμβαστική τροπολογία. Διαφωνώ δεν θεωρώ ότι καλύπτονται και γιατί να μην τις ψηφίσουμε ξεχωριστά αντί αυτή η περιπτώση. Πολύ ωραία, γιατί όχι, ε, πράγματι τα ψηφίσουμε ξεχωριστά. Πολύ ωραία, ψηφίζουμε λοιπόν ε, τροπολογία υπαριθμών 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται. Νομίζω εδώ πρέπει να έχουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ για την τροπολογία υπαριθμών 32. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. 35 υπέρ, θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν ε, βοηθούσαν λιγάκι οι συντονιστές. Η τροπολογία 33 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 40 αποσύρθηκε. Η τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Εις 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. η 34 και 53. Ε, πάμε τώρα στην συμβαστική υπαριθμών 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή η συμβιβαστική 51 υπέρ, μα, με συγχωρείτε, η τροπολογία 51 υπέρ κατά αποχές, εδώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Ich ε, schließe die Abstimmung. Έκλεισε η ψηφοφορία. 32 υπέρ δεκτή. Η 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή ή 55 υπέρ κατά αποχές. Αυτό πρέπει να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επανήθευση για την 54 παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. 23 υπέρ, η 57 ε, υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 59 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 67 τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 69 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επανλήθευση για την 71. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Δεκτή. Η 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η συμβαστική 15 74 ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή. Η τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Η 81 υπέρ κατά αποχές. Δε... Απορρίπτεται. Η 82 υπέρ κατά αποχές Πάμε στην 84 ε, ε, υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 87 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω πρέπει να το ελέγξουμε ηλεκτρονική επαλήθευση 88 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η 89 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 16, η συμβαστική 16 υπέρ κατά Η 17 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η τροπολογία 102 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η τροπολογία 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 104 ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε παρακαλώ Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 109. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά απορρίπτεται η 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή ή 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 127 υπέρ κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 129 Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή και περνάμε τώρα στην ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ Έκλεισε η ψηφοφορία. Δεκτή η πολιτική ανταγωνισμού. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια της γνωμοδότησης. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ε, ψηφοφορία για την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του 2018 και εκεί ε, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο εισηγητή επιθυμεί το λόγο, ο συνάδελφο Αρακόβατ. Σα ευχαριστώ. Έχω δύο σχόλια προ το παρόν. Νομίζω ότι οι τροπολογίε ήταν ισορροπημένε και καταφέραμε το μήνυμά μα να είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. Ε, η συμβιβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η συμβιβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Για την τροπολογία 13 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική η 6. Η 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 30 η τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η τροπολογία 38. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 38. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 25 με 17 είναι το αποτέλεσμα. Επόμενο. Η συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, ε, δεκτή. Η, με η τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή. Η συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και έτσι λοιπόν πάμε τώρα στην ε, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έκλεισε η ψηφοφορία. Και εδώ ε, θερμά στον εισηγητή. Άρα ε, φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το σημείο 8, παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κατεξουσιοδότησης πράξης σχετικά με τη δέσμη ευελιξίας για τα προγράμματα προώθησης του ίνου. Έρχεται η Κομισιόν. Thank you, Mr. Uh, President. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το συγκεκριμένο σημείο χρονολογείται από ένα ψήφισμα του ίδιου του Κοινοβουλίου σε σχέση με τη δασμολογικά μέτρα που ε, επέβαλαν οι ΙΠΑ μετά από τα απορίσματα του ΠΟΕ ε, σε σχέση με την υπόθεση Boeing Airbus. Έχουμε λοιπόν ψήφισμα τη ΣΥΝΤΑ. Το Κοινοβούλιο ε, υιοθέτησε διάφορες ε, κατευθύντριες γραμμές και προσανατολισμού για να ζητήσει από την Κομισιόν να στηρίξει τον τομέα του κρασιού ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτές τους δασμούς. Υπάρχει μια μακρά ιστορία πίσω από την διαφορά στον ΠΟΕ. Πάντως παραμένει γεγονός ότι τα μέτρα που υιοθέτησαν οι ΙΠΑ εγκρίθηκαν από τον ΠΟΕ. Είναι ατυχές ότι επέλεξαν συγκεκριμένα ε, ε, γεωργοτροφημικά προϊόντα, αλλά αυτή είναι μια τάση που είδαμε και στο παρελθόν όταν πρόκειται για ζητήματα εμπορίου. Όταν η Ευρώπη είναι ο στόχος, ο, κατε, στόχος είναι τα γεωργικά προϊόντα. Περισμένο παράδειγμα είναι το ρωσικό εμπάργο. Ε, είναι ε, περίεργο και η Κομισιόν επαλημένα έχει πει ε, ότι θέλει να διαπραγματευτεί λύση με τις ΗΠΑ σε σχέση με την μακρά, μακρά αυτή εμπορική διένεξη. Εν πάση περιπτώσει και σε αυτό το πλαίσιο και μιλώντας ειδικά για τον Ίνο, τα μέτρα των ΙΠΑ είναι περιορισμένα ε, στον γενικό του πεδίο ορίζουν δηλαδή τους δασμούς σε ένα επίπεδο 25% για το κρασί για τέσσερα, τέσσερις χώρες, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει αναφερθεί η ιδέα ότι αυτοί οι δεσμοί προβλέπονταν και φόβος μας ήταν ότι θα επεκτείνονταν σε όλα τα προϊόντα ίνου και στους αφρόδεις ίνους ε, και για όλα τα κρατη και ότι μπορεί να επιβάλλονταν σε πολύ ψηλότερο επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο 100%. Δεν είναι παρηγοριά βέβαια για αυτό το τομέα και για τον αντίκτυπο στα κρατη ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχα χειρότερα η Κομισιόν προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα επιδεινωθούν άλλο. Και στο πλαίσιο αυτό έπρεπε να έχουμε υπόψη μας ε, τις παράλληλες απειλές από πλευράς ΗΠΑ για επιβολή δασμών σε σχέση με εισαγωγές Ίνου και Αφρόδου Ίνου από την Γαλλία ως ε, αντίπεινα για τον ε, φόρο για τις ψηφιακές πωλήσει. Η Κομισιόν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θα δείξει πλήρη ελεγγύη με τη Γαλλία και με τα άλλα τα κράτη-μέλη όσον αφορά αυτές τις διμερείς ε, απειλές. Έχουμε κάποια καλά νέα γιατί εντωμεταξύ οι διαπραγματεύσει σε διμερές επίπεδο στη Γαλλία οδήγησαν στην αποφυγή ε, ύπαρξη αυτού του κινδύνου και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ε, λύση και στο θέμα του φόρου ψηφιακών πωλήσεων. Το ψήφισμα λοιπόν έχει ψηφιστεί τον Νοέμβριο και ζητά από την Κομισιόν να λάβει μέτρα για να στηρίξει τον τομέα του Ίνου και η Κομισιόν απάντησε με τρεις συγκεκριμένους κανονισμούς. Ένας εξ αυτών είναι μία κατεξοδότηση πράξη, ένας κανονισμός κατεξοδότηση πράξης με τρία συστατικά. Το ένα είναι να αρθεί ο πενταετής περιορισμός για τη λειτουργία των προγραμμάτων, πράγμα που θα βοηθήσει τους φορείς να παγιώσουν τις ε, στοχευμένες αγορές και να αφήσουν τους κύκλους εργασιών να, περάσουν, να ισχύσουν για τα πέντε χρόνια μέχρι το τέλος του προγραμματισμού τον Οκτώβριο δηλαδή του 2023. Ε, δεύτερο σκέλος είναι ότι επιτρέπεται οι φορείς να αλλάξουν τις αγορές προορισμούς. Για παράδειγμα, ε, μπορεί κάποιος να θελήσει να περικόψει να σταματήσει τις δραστηριότητε πρόθεσης σε ένα συγκεκριμένο κράτος, ας πούμε στη ΣΥΠΑ, και να τις στρέψει σε άλλες πιθανές αγορές ε, όπως ε, η Κίνα, ο Καναδάς, η Αυστραλία και ούτω καθεξής. Και ένα άλλο μέτρο το οποίο εισάγει βελτιωμένη, μάλλον αυξημένη ευελιξία στην περίπτωση που οι, ε, οι νοπαραγωγοί αλλάξουν τον προορισμό και τον προορισμό στόχο, τότε θα υποστηρίξουμε ε, τους στόχους και για τις υπάρχουσες δραστηριότητες, δηλαδή δεν θα υποστούν καμία οικονομική αλλαγή σε σχέση με την αλλαγή αυτών των στόχων. Μετά έχουμε δύο εφαρμοστικούς κανονισμούς παράλληλα. Ο ένας επιβάλλει στην Κομισιόν να αυξήσει το ρυθμό και το ποσοστό μάλλον χρηματοδότησης των μέτρων πρόθεσης από το 50% που ισχύει ε, θα ανέλθει στο 60% και ο δεύτερος ε, προσφέρει την ευελιξία ώστε τα μέτρα προώθησης θα μπορούν να προσαρμοστούν ε, αρκετές φορές μέσα στον ίδιο χρόνο και όχι μόνο κάθε δύο χρόνια όπως προβλέπεται μέχρι τώρα. Λόγω του επίγοντος χαρακτήρα και της ευαισθησίας αυτών των μέτρων δουλέψαμε σκληρά ώστε να εισαχθούν όσο γίνεται πιο σύντομα και παρουσιάστηκαν ήδη στα κράτη-μέλη στην ε, ε, ε, Επιτροπή που ασχολείται με το κρασί στις 15 Ιανουαρίου ήδη τον, και γκρίθηκαν και θα ε, περάσουν και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από τις ε, φυσιολογικές δραστηριότητες, ε, προθεσμίες με συγχωρείτε, ε, όσον αφορά την προθεσμία ελέγχου και εξέτασης κτλ. Τα μέτρα έχουν ήδη ανακοινωθεί στα κράτη-μέλη και στους ενδιαφερόμενους, οπότε ήδη δουλεύουν προβλέποντας αυτά τα μέτρα και με βάση αυτή την αυξημένη ευελιξία ε, θα μπορέσουμε έτσι να περικόψουμε σε κάποιο βαθμό τον αντίκτυπο των δασμολογικών μέτρων των ΙΠΑ. Τελικά όμως η πραγματική λύση σε αυτά τα σφραγμούς είναι η άρση των, μέτρων, των δασμολογικών μέτρων. Ο Επίτροπος ήταν στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα, θα ξαναπάει μέσα στις επόμενες εβδομάδες γιατί είναι μεγάλη προτεραιότητα στην ατζέντα του και εμείς θα, κάνουμε, θα βάλουμε κάθε λογική προσπάθεια ε, με τα κρατη ώστε να ε, αρθούν αυτά τα μέτρα όσο γίνεται πιο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή που μας κάνατε. Ε, έχουμε βέβαια κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε. Δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ε, τηρήσετε το ένα λεπτό. Συνάδελφος Αγγιλάρ. Ευχαριστώ. Τα νέα μέτρα προώθησης του ίνου είναι ευπρόσδεκτα, αλλά δυστυχώς είναι ανεπαρκή. Ε, ο τομέας αυτός έχει πληγεί ε, από την επιβολή δεσμών από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν αρκεί αυτό το μέτρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο προορισμός των 40% των αμπελονικών μα ε, προϊόντων. Οπότε ε, καλή πρόθεση, αλλά είναι πιο μακροπρόθεσμο μέτρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι βραχυπρόθεσμη λύση για να βελτιωθεί η κατάσταση ή να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες προς τους Ευρωπαίους και κυρίους Ισπανούς αμπελουργούς. Καμία αγορά δεν ανοίγει από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν θέλουμε βαλωματικά μέτρα, αλλά πιο αποτελεσματικέ λύσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να κοφεύει στις εύλογες ε, απαιτήσει ενός κλάδου που εξακολουθεί να νιώθει από περιθωριοποιημένος από τις προτάσεις και η μόνη λύση που προτείνεται είναι κάποια μέτρα προώθησης παραγωγής παραγωγής. Ευχαριστούμε πολύ. Οι διερμηνείς μου επισήμων ότι πρέπει να μιλάτε πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε πάλι για δασμούς. Διζητήσαμε ε, την βοήθεια προς τον πελοϊνοπαραγωγικό ε, τομέα και όντως ε, κάνετε αυτά τα πρώτα, μέτρα που δεν αρκούν. Ελπίζουμε όμως ε, πως θα συνεχίσουν να ισχύουν πάνω από πέντε χρόνια για να ενισχυθεί η ισχύ τους. Γιατί στην Ευρώπη και στη Γαλλία κυρίως έχουμε αριστεία στον τομέα αυτό και πρέπει να το προστατεύσουμε. Δεν θα πρέπει όμως ούτε και να αγγίξουμε τα στάνταρ ασφάλειας ε, για τα προϊόντα τράφημα, γιατί ο Χόγκαν στη Γόσικτον μίλησε για εξάλληψη φραγμών, ε, κατάργηση μάλλον φραγμών στον τομέα ε, των τροφίμων. Εμείς είμαστε ωστόσο δεσμευμένοι να διατηρήσουμε το καλύτερο για τους παραγωγούς μας και για τους καταναλωτές μας και κυρίως στο γεωργικό τομέα δεν πρέπει ποτέ το ξεχνάμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεκάστρο. Ναι, εγώ έχω να κάνω κάποιες ε, αναφορές. Καταρχάς, ένα ευχαριστώ στην Κομισιόν που ενέκρινε αυτή τη σημαντική κατεξοδότηση πράξη. Όπως ξέρετε, εμείς οι συντονιστές υπερψηφίσαμε να μπει στην γρήγορη διαδικασία, ακριβώ για να μπορέσει να εφαρμοστεί γρήγορα. Ευχαριστούμε λοιπόν γι' αυτό. Τώρα, για το μέλλον, θα ήθελα να πω τα εξή. Όταν γίνεται λόγος για το άρθρο που αφορά τα πέντε χρόνια, γίνεται αναφορά στο ότι πρέπει να αιτιολογηθούν ε, ευρέω, αν ε, αυτό παραταθεί για πάνω από πέντε χρόνια. Εγώ πιστεύω πω θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε στο μέλλον γιατί διαφορετικά θα ήταν αυτό ένα γραφειοκρατικός φόρτο. και το ίδιο και σε αφορά το άρθρο 2 νομίζω ότι είναι που αναφέρεται στα αίτια ε, νοτέρα βία που εμποδίζουν την ολοκλήρωση ενό προγράμματο. Είναι προφανέ ότι αν υπάρχει νοτέρα βία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Οπότε αυτό θα ζημιώνει τους παραγωγούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας είπατε. Για μας, για την ομάδα Renew, αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, και νομίζω το κατασέμε σαφές τον Νοέμβρη στο ψηφισμά μας. Η κατάσταση των εινοπαραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βελτιωθεί και τώρα μας παρουσιάσετε τα συγκεκριμένα μέτρα. Εγώ πιστεύω ότι αυτά θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε. Τώρα, κατά πόσον θα αρκούν, αυτό θα το δούμε. Για μένα που έχει σημασία είναι ότι θα υπάρχει μια ταχεία διαδικασία στις 29 πρώτου. Ε, θα ξεκινήσουμε με την εφαρμογή αυτών των μέτρων και κατόπιν όλα αυτά θα γίνουν αισθητά στους ε, παραγωγούς. Τώρα, κατά πόσον ε, αυτά τα εργαλεία κρίσης που έχουμε θα πρέπει να επεκταθούν ή όχι, αυτό νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινή γεωρικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Καταρχά, ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κατεξουσιοδότηση κανονισμό για να φέρει μεγαλύτερη ελαστικότητα στην προώθηση ε, του ίνου. 25% δασμός ε, στα μπελονικά προϊόντα εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών ε, κατέφερε σοβαρότατο πλήγμα σε χιλιάδες παραγωγούς και αμπελουργούς. Ήταν πολύ ισχυρό πλήγμα για τον αμπελοϊνικό τομέα σε πολλέ χώρε, όπω και στην Ισπανία. Οπότε ήταν απαραίτητο να αντιδράσουμε και να δώσουμε ένα ελάχιστο περιθώριο λιγμών ώστε οι εξαγωγεί να μπορέσουν να αναπροσανατολίσουν τα προϊόντα του και να τα προωθήσουν σε άλλε αγορέ. Με τον κατεξοδότηση κανονισμού, ε, ακολουθούμε μια σωστή πορεία. Θα πρέπει όμως να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία ώστε τα μέτρα που θεσπίσαμε να τεθούν σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατό αλλά έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μα. Γιατί δεν αρκούν κάποιες βραχυπρόθεσμε εμβαλωματικέ λύσεις. Θα πρέπει να έχουμε κατεπηγόντω διαπραγματεύσεις για να τεθεί επιτέλου ένα τέρμα στους δασμούς σε όλα τα αγροδιατροφικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η κατάλληλη λύση για τους γεωργούς κτηνοτρόφου αλλά και για τον αμπελοϊνικό μα τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Αγγιλέρα. Ευχαριστώ. Για τον κανονισμό αυτό, όπως και οι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι καλή η πρόθεση, αλλά κακή η πρόταση. Γιατί ουσιαστικά αφαιρεί ε, κονδύλια από άλλα επενδυτικά προγράμματα και τα προσανατολίζει στην προώθηση, στην προαγωγή των προϊόντων. Και με τον κόλαφο αυτό που έλαβαν οι αμπελουργοί δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε μία πρόθεση που μάλιστα απορροφά κονδύλια από άλλα επενδυτικά προγράμματα που έχουν ήδη σχεδιαστεί. Παίρνουμε από το ένα και δίνουμε στον άλλο. Αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και πάλι. Και μπορεί να είναι καλά εστιασμένο το μέτρο και αν χρηματοδοτείται με χρήμα, έχει καλός. Αν όμως ε, ε, προσπαθούμε να αντισταθμίσουμε το, το πλήγμα που υπέστησαν από τους δασμούς, θα πρέπει να βρούμε κονδύλια καινούρια και όχι μεταφορά από άλλους τομείς. Ευχαριστώ κύριο Διτό, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά Νομίζω ότι αντιμετωπίζει το θέμα σαν να είναι συγκυριακό, ενώ είναι διαρθρωτικό. Γιατί σε θέματα ηλεκτρονικών, αυτοκινητοβιομηχανίας, αεροναυπηγικής, ε, δυστυχώς πολύ συχνά η γεωργία είναι το αντάλλαγμα στις ε, διεθνείς συμφωνίες και θυσιάζεται στο βομάλων άλλων προϊόντων. Καλή πρόθεση των γεωργικών προϊόντων, αλλά δεν αρκεί δεν αρκεί αυτή η διαφήμιση και η πραγωγή που κάνουμε. Και όπως είπαμε και τον Αύριο, πιστεύω ότι μπορούμε να κινητοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Γιατί σε καταστάσεις που σήμερα μας παρουσιάζεται ως συγκυριακές, αλλά στην ουσία είναι διαρθρωτικές, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη συμπαράσταση όταν εμφανίζονται τέτοιες περιστάσεις ε, στην αγορά. Και θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια. Γιατί να μην κινητοποιήσουμε λοιπόν και για τη Γεωργία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ κύριος Ντόρφμαν. Ähm, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συμφωνώ με όλους αυτούς που είπαν ε, πριν από μένα ότι βεβαίως ε, και είναι πολύ καλά τα μέτρα, αλλά είναι απλά σταγόνο το ωκεανό. Και όπως είπαν και οι προραλήσαντες, ε, επειδή οι γεωργοί είναι εκείνοι που καλούνται να λύσουν τα προβλήματα που προκάλεσε η προκάλεσαν οι αεροπορικέ μεταφορές, νομίζω ότι πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα για να τους βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τους δασμούς, το Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου αυτή τη στιγμή ερευνά το θέμα των δασμών, τα 6,5 δι ευρώ τα οποία εγκρίθηκαν ε, δεν μπορούν να επιτευχθούν με δασμούς και γι' αυτό λοιπόν αναφέρεται ότι νέα προϊόντα σε κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβαρύνονται με νέου δασμού στην Ιταλία το κρασί δεν επιβαρύνεται, αλλά υπάρχει ο φόβος ε, στο μέλλον να αυξηθούν οι φόροι μέχρι και κατά 100%. Ε, πολλοί μου λένε ότι εδώ και καιρό οι εισαγωγεί δεν έχουν παραγγείλει ούτε, μία, ούτε ένα μπουκάλι, γιατί φοβούνται ότι τελικά ε, θα τους αναγκάσουν να πληρώσουν δασμούς. Δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω, ξέρετε να υπάρχει κάτι καινούριο και από το ταξίδι του Επιτρόπου, κάτι που να αφορά στο μέλλον, τι θα γίνει, τουλάχιστον να μην επιδεινωθεί η κατάσταση σε σχέση με αυτή που ισχύει τώρα. Συνάδελφος Σάντερ. Ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις Βέβαια, έχει παραμείνει κάτι εκρεμές. Μας είπατε για την ενεργοποίηση των μηχανισμών της κοινή οργάνωσης αγοράς και τη θέσπιση κάποιων μέτρων αντιστάθμισης των τομέων που έχουν πληγεί. Από αυτή την άποψη όμως οι προτάσεις δεν λένε τίποτα. Θα ήθελα η Γενική Διεύθυνση Άγκρη να ανασκομποθεί και να εισακούσει τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ε, προέχει ε, τα κείμενα αυτά να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Και θα ήθελα να προτείνω και στους συντονιστές να εγκύψουν σε αυτό το θέμα και ενδεχομένως ε, να εκπονήσουν και ένα ψηφισμά για την αντίρρηση. Ευχαριστώ εκ μέρους του Ευρωπαίων και δι των ε, Γάλλων αμπελουργών που έχουν πληγεί από τους Αμερικανικούς δασμούς. Ευχαριστώ κύριε Σαντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω τα επίγοντα αυτά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ με το περιεχόμενο των μέτρων, αν και συμφωνώ με τους συναδέλφους ότι είναι ανεπαρκή για να αποφύγουν ή να αποτρέψουν μια επιδείνωση της κατάστασης στον αμπελονικό κλάδο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις, γιατί ε, Προσπαθείτε να δώσετε απάντηση με συγκυριακά μέτρα σε ένα διαρθρωτικό πρόβλημα. Μην το ξεχνούμε αυτό. Επίσης, πώς θα, πώς θα χρηματοδοτήσουμε. Ε, γιατί θα χρειαστεί συμπληρωματικά κονδύλια. Με ένα πό θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Πώς θα χρηματοδοτήσετε λοιπόν την εκτέλεση που περιλαμβάνει που ε, χρηματοδότησε από 50 σε 65% και για τα διαρθρωτικά θέματα δεν, θα έχουμε, δεν χρειάζονται και κάποια μέτρα αγορά για να αντιμετωπίσουμε τέτοιε κρίσει τη στιγμή που επεξεργαζόμαστε την αναθεώρηση τη ΚΑΠ και δι τη κοινή οργάνωση αγορά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω, μου είπαν και πάλι ότι ε, δεν πρέπει να μιλάτε τόσο γρήγορα για να μπορούν και οι συνάδελφοι να ε, έχουν το χρόνο να μεταφράσουν σωστά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ έχω μία ερώτηση γιατί πάρα πολλά ελέγχθησαν ήδη ε, σε σχέση με τα διαρθρωτικά προβλήματα. Πάνω από ένα δις ευρώ δαπανούμε για την πρόθεση πωλήσεων του κρασιού. Έχουμε τώρα την Πράσινη Συμφωνία. Έχουμε ε, κλιματική κρίση. Ε, πρέπει να εργαζόμεθα ε, με βάση την βιωσιμότητα. Αλλά τα μέσα ενημέρωση λένε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες εποφελούνται από αυτά που ισχύουν σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν γνωρίζετε ποια είναι τα αντίμετρα που μπορούμε να λάβουμε. Γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να απειληθούν με την υποστήριξη των περιφερειακών ε, πωλήσεων. Όπως είπε και η κυρία Αγγιλέρα, τα χρήματα αυτά μπορούμε ε, ενδεχομένως ε, να τα κλέψουμε από άλλα προγράμματα για να κλείσουμε το κενό, αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε τους μικρούς ε, γεωργούς και ενοπαραγωγούς και όχι αυτές τις πολυεθνικές που τις χρηματοδοτούμε και από πάνω. Συνάδελφος Τολερέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έλαβε υπόψη το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλαβε τις σχετικές δράσεις. Νομίζω ότι ε, ευτυχώς σπεύσαμε και κινηθήκαμε και μάλιστα υπερκομματικά. Ευχαριστούμε για το κείμενο, αν και θα περιμέναμε πιο φιλόδοξες προτάσεις πέραν αυτής της ε, επίγουσης διαδικασίας. Και έχουμε κάποιους παραγωγούς που είναι στο πιο μεγάλες, αλλά έχουμε και μερικές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που κινδυνεύουν με πτώχευση. Και είναι κρίμα να έχουν προσπαθήσει τόσα χρόνια να διεισδύσουν στην Αμερικανική αγορά οι Ευρωπαίοι παραγωγή και να έχουμε κάποιες μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, όχι πολυεθνικές που ήδη έχουν ε, οργανωθεί, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις να απειλούνται με πτώχευση. Ανεπαρκή λοιπόν είναι τα μέτρα, παρόλο που είναι ευπρόσδεκτα ε, και θα πρέπει να Προτείνουμε και μέτρα της αγοράς και ένα ταμείο αντιστάθμισης, αποζημίωσης. Και ήδη από το Φεβρουάριο φαίνεται ότι αρχίζει ένα σπιράλ. Ε, έχετε προβλέψει δημο... διπλωματικά μέτρα για να αποφύγετε αυτή τη δαμόκλειο σπάθη που επικρεμάται πάνω από τους γεωργούς. Επίσης, ε, δεν μπορούμε να επισπεύσουμε τη λήψη των μέτρων, ώστε σε παρόμοιες κρίσεις στο μέρο να δρούμε πιο τάχιστα. Ευχαριστώ κύριε Ρίτσι. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα, δύο δευτερόλεπτα θα μιλήσω ακόμα. Εγώ πιστεύω πως υποφέρουμε από τους δασμολογικούς πολέμους. Έχουμε επιβάλει ε, δασμούς στη ΣΥΠΑ και θα ήθελα η Κομισιόν να σκεφτεί την άρση αυτών των δασμών και μιλώ ειδικά για το σκοτσέζικο ουίσκι που είναι τόσο σημαντικό για μας και να ε, επιτρέψει έτσι και στη ΣΥΠΑ να αποσύρει τους δικούς δασμούς. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Έθελα λοιπόν να δώσω το λόγο ε, στον ε, εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν έχει την καλοσύνη να είστε πάρα πολύ σύντομος γιατί ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρονικό διάστημα που προβλεπόταν για αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που εθίγησαν είναι το επίπεδο παρέμβαση τη Κομισιόν για να στηριχθούν οι παραγωγοί. Και στο πλαίσιο αυτό, ε, να πω στον κύριο Ανδρίο καταρχά ότι είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα ότι αυξάνουμε ε, την συμβολή από το 50% στο 60%. Ε, υπάρχει όμως ε, υποδαπάνη σε πολλά κράτη-μέλη. Τα χρήματα υπάρχουν. Είναι πιεστική ανάγκη αυτή τη στιγμή. Τα χρειάζονται οι παραγωγοί. Τώρα, η συμβολή της Κομισιόν που θα αυξηθεί στο 60% μέχρι ένα γενικό ανώτερο όριο του 80%. Υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη ε, για περισσότερα χρήματα για να βοηθηθεί ο τομέας. Η άλλη ερώτηση αφορούσε τον φόβο των παραγωγών ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε κλιμάκωση. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θέλουμε να αποφύγουμε ένα τέτοιο σενάριο όπου δηλαδή οι ΙΠΑ θα ε, επιβάλλουν δασμούς μέχρι και 100%. Κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό, το ανέφερα ήδη. και ανέφερα και τις συζητήσεις μεταξύ του Τραμπ και του Μακρόν για την επιβολή του ψηφιακού φόρου. Αλλά ένα από τα σαφή μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι εάν δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τον αντίκτυπο επιτόπου, για αυτούς τους δεδομένους που έχουν εφαρμοστεί σήμερα, αυτό που θέλω να αποφύγω σε πάση θυσία είναι να ε, επικρατήσει πανικό στον τομέα αυτό, γιατί το κρασί είναι πολύ σημαντικό προϊόν και το περισσότερο, η περισσότερη παραγωγή καταναλώνεται εδώ στην Ευρώπη. Εάν υπάρξει λοιπόν αντίληψη στην αγορά ότι η κατάσταση θα χειροτρέψει, πολλοί κόσμος ή ε, εστιατόρια ή ε, έμποροι μπορεί να περιμένουν να αγοράσουν μέχρι να του πέσουν οι τιμές. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν να μην, να μην περάσει το μήνυμα ότι ο τομέα περνά κρίση. Πρέπει να τετρίσουμε την ψυχραιμία μας. Και αυτό που θα πω τώρα το είναι πολύ σημαντικό επίσης. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε αυτά τα μέτρα να αρθούν. Όχι να μην υπάρξει κλιμάκωση, αλλά να καταργηθούν και τελείως. Εμεί έχουμε πει επανειλημμένα πω οι δασμοί δεν είναι λύση ε, για αυτές τις εμπορικές ενέξει. Πρέπει να βρούμε διαπραγματεύσεις ε, λύσεις και τα ζητήματα να ρυθμίζονται εύκολα. Α πούμε εδώ στη ΣΥΠΑ να αποσύρουμε ε, δασμού για τη ΣΥΠΑ ώστε να του ενθαρρύνουμε να δράσουν και αυτοί αντίστοιχα. Έχετε υπόψη ότι οι δικοί μας δασμοί ήταν άμεση αντίπεινα για αυτό που έκαναν εκείνοι πρώτοι. Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι το Μάιο-Ιούνιο έχουμε ΠΟΕ για την και απόφαση για την ε, υπόθεση Boeing, πράγμα που θα μας επιτρέψει εμείς να επιβάλλουμε δασμούς ε, σε προϊόντα των ΗΠΑ. Δεν είναι κάτι που θέλουμε ή επιθυμούμε να κάνουμε, αλλά η Κομισιόν έχει πει ότι δεν θα διστάσει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των δικών μας παραγωγών, είναι παραγωγών και όλων των παραγωγών. Και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτοί οι δασμοί έχουν επιβληθεί όχι μόνο στον τομέα του κρασιού, αλλά και στο πνευματόδη, στο ε, ελαιόλαδο, στα γαλακτοκομικά, στα τυριά και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι παραγωγοί και άλλοι τομείς της γεωργικής μας κοινότητας που πλήττονται αυτή τη στιγμή και είναι προς τιμή του, φορέα, του, κλάδου του κρασιού και είναι επιτυχής ιστορία των τελευταίων ετών. Οι εξαγωγές μας πάνε πάρα πολύ καλά. 12 δις ευρώ ε, σε προϊόντα κρασιού εξάγουμε και προς τη ΣΥΠΑ. Και γι' αυτό και μας στόχευσαν με αυτό το προϊόν, γιατί θέλουμε, θέλουν να μας χτυπήσουν σε έναν τομέα επιτυχή. Και κλείνω. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και αρκετοί το αναφέρατε ότι πολλή ζημιά γίνεται επίση στι ίδιε τι ΗΠΑ. Διότι τα ευρωπαϊκά κρασιά είναι πολύ δημοφιλή για του Αμερικανούς καταναλωτέ. Υπάρχει ολόκληρη ροσκλάδο εισαγωγή. οι αποθήκε, τα εστιατόρια, οι έμποροι. Αυτοί βγάζουν λεφτά από τα ευρωπαϊκά κρασιά. Και γι' αυτό και μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου έγραψαν στον πρόεδρο Τραμπ και εξέφρασαν ε, πολύ έντονε αντιρρήσει για αυτές τις αποφάσεις του. Ελπίζουμε λοιπόν πως κάπω θα εισακωστούμε στους εμπορικού κύκλους ώστε να αυτό ίσως να εξηγεί και γιατί δεν κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο η κατάσταση γιατί οι δασμοί βλάπτουν και τις δύο του Ατλαντικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε σύντομοι όμως. Πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Το 10% αύξηση για την προώθηση δεν είναι φρέσκο χρήμα. Είναι χρήματα που υπάρχουν στα κρατημέλη και που προβλέπονται για μέτρα και προγράμματα για επενδύσει που ήδη έχουν προγραμματιστεί. Δεν είναι χρήματα που δεν έχουν δαπανηθεί. Αυτό είναι ψέμα. Είναι χρήματα για, ε, χρήματα για προγράμματα για ε, επενδύσει που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Δηλαδή, βγάζουμε από το ένα σακούλι και τα βάζουμε στα άλλα. Έχει θετικά στοιχεία, αλλά δεν πρόκειται για φρέσκο χρήμα. Είναι χρήματα που πάνε από αλλού στον τομέα του κρασιού. Θέλετε να απαντήσετε. Αν νόμιζα πως το είπα αυτό, ε, γιατί τόνισα και αυτό περιλαμβάνει και την Ισπανία. Υπάρχει σημαντική υποδαπάνη των εθνικών προγραμμάτων ε, στήριξης ε, και ο Πίτροπος Χόγκαν ήταν στη Νέα Υόρκη πριν από λίγο καιρό και έκανε αυτή την παρατήρηση στους Ισπανούς εταίρους του ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να απορροφήσουν τα χρήματα που είχαν προβληθεί. Τα χρήματα υπάρχουν. Είτε δαπανώνται για επενδύσεις, είτε πρόκειται για την ε, μείωση των τιμών κτλ. Η προώθηση είναι επιλογή των κρατών μελών. Αλλά τώρα έχουν προσανατολισμό ότι πρέπει να εστιάσουν τι προσπάθειέ του στην προώθηση και γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μα ότι η Ισπανία. έχει τη δυνατότητα να βάλει τα υπόλοιπα λεφτά μέχρι το ανώτατο όριο το 80% χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Διευθυντά για αυτές τις ε, πληροφορίες. Ε, σίγουρα ε, θα παραμείνουμε σε επαφή. Ε, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες επιθυμίες εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, κλείνει το επίσημο κομμάτι της σημερινής, του σημερινού πρωινού και θα ξεκινήσουμε τώρα με τον επίσημο κομμάτι με τους συντονιστές. Οι υπόλοιποι θα τα πούμε εδώ στις 2.30 με πρώτο θέμα την υγεία των ζώων. Ευχαριστώ πολύ.